αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε σιγά σιγά γιατί είναι φορτωμένη η ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί. Θα ξαναρχίσουμε, θα αρχίσουμε μάλλον το διαρθρωμένο διάλογο με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, τον κύριο Τιτιέ Ρέντερς, και θα ακούσουμε και παρουσιάσεις από τους αρμόδιους υπουργούς για θέματα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας από την κρατική προεδρία που ασκεί αυτό το καιρό την προεδρία στο Συμβούλιο. Αρχίζουμε όμως τη σημερινή συνεδρίαση με το σημείο 7 για την πρόσληψη διάδοσης ε, τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα για μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από την περασμένη σύνοδο Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Μάλλον κατά τη διάρκεια την περασμένη Τρίτη είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο Γιωχάνσον. Έχει δείχνει σε εμπλοκή αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διαπραγματευτική του εντολή και το Συμβούλιο. Αλλά η Επίτροπος Γιωχάνσον επιτέλους δεσμεύτηκε να φέρει συμβιβαστικέ προτάσεις. τις οποίες συστηματικά και επίμονα ζητεί η Επιτροπή μας. Πριν από τις τεχνικές συνεδριάσεις θα φέρει συμβιβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις. Και τελικά να απεμπλακεί αυτό το ζήτημα Όπως γνωρίζετε, η κατάσταση έχει ως Το, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το θέμα αυτό στην περασμένη ακόμα θητεία, σε πρώτη ανάγνωση. Εμείς ξεκινήσαμε, αλλά το Δεκέμβριο του 2019 η Επιτροπή μας ψήφισε για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Με στόχο να βρούμε μια δεύτερη συμφωνία. Έχουν γίνει πολιτικοί τριμερείς διάλογοι, τρεις στον αριθμό, κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Με μηδενικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε τον εισηγητή μας τον κύριο Γιάκη της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για να μας πει πώς έχει η κατάσταση στον διοργανικό διάλογο και διαπραγματεύσεις. Και μετά ε, θα γίνει και μια συζήτηση, θα μιλήσουν πρώτα οι σκιώδεις ηγητές με τη σειρά. Ας ακούσουμε πρώτα όμως τον εισηγητή μας. Κύριε Γιάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα περάσω τώρα στα πολωνικά. Korzystając z e, mandatu przyznanego przez e, Wysoką Komisję 17 października zeszłego Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 17 Οκτωβρίου μας έδωσε διαπραγματευτική εντολή και μαζί με τους άλλους συναδελφούς της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ αρχίσαμε τη σκληρή δουλειά. Μέσα σε ένα τρίμηνο σχεδόν είχαμε 16 παρακαλώ συναντήσεις, 7 τεχνικής φύσεως τρεις ε, τριμερούς διαλόγους. Ε, ε, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα έγγραφα του Κοινοβουλίου από εκείνα του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση επιλέξει από το Συμβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλα αυτά και χάρη στη σκληρή δουλειά όλων των ε, βουλευτών, επιτύχαμε πολλά. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος έγινε το Δεκέμβριο. Ορίσαμε τι εστί τρομοκρατικό περιεχόμενο και ποιες είναι αξιόπινες πράξεις. Μιλήσαμε για τα φίλτρα στο διαδίκτυο, μιλήσαμε και για την εντολή απομάκρυνσης αυτού του περιεχομένου από το διαδίκτυο. Σημαντικά άρθρα ήταν το 7, το 10, το 16 όλα αυτά είναι νομικά ζητήματα και υπάρχει και άρθρο για την αξιολόγηση. Ε, υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί ε, που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης. Την Τετάρτη η κυρία Κάλιου Ραντ και ο κύριος Μπράιερ διοργανώνουν μία συνάντηση με εμπειρογνώμονες. Στο Φλεβάρι θα δούμε την Ευρωπόλ και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σας προσκαλώ για σας. Είμαι βέβαιος ότι και αυτά τα πάνελ των εμπειρογνωμόνων θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή πάντως θα πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι το έγγραφο δεν έχει τεχνικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημεία διαφωνίας και τριβής σε δύο σημεία, όπως σας είπα, διαφέρει πάρα πολύ η προσέγγιση του Κοινοβουλίου από εκείνη της Επιτροπής ε, και του Συμβουλίου. Το πιο επίμαχο είναι οι εντολές απομάκρυνσης του περιεχομένου αυτού του τρομοκρατικού από το διαδίκτυο και μάλιστα διασυνοριακά. Εκεί αντέδρασαν ε, με πολύ μεγάλη σφοδρότητα οι εταιρείε ε, ε, παροχής ε, υπηρεσιών διαδικτύου. Το Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι κινδυνεύει η ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο. Έχω συχνές επαφές και συναντήσεις με πολλούς εκπροσώπους των άλλων πολιτικών ομάδων και ξέρω ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε σε αυτά που απαιτεί το Συμβούλιο. Επίσης γίνεται λόγος για αυτόματα φίλτρα ελέγχου στο ίντερνετ και αυτό είναι επίμαχο ε, και αμφιλεγόμενο θέλει ε, το Συμβούλιο να προτείνει κάποια συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία εμείς έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε πιο αυστηρή νομοθεσία γιατί αυτό απειλεί την ελευθερία του διαδικτύου. Θέλω να πω συνοψίζοντα ότι έχουμε πετύχει ήδη πάρα πολλά με αυτό το κείμενο, απομένουν αυτά τα δύο τα οποία όμως είναι βασικά και κομβικά και πρέπει να λυθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διαφυλάξει και να υπερασπιστεί την ελευθερία της έκφρασης στο ίντερνετ, το Συμβούλιο θέλει να χρησιμοποιήσει τα νέα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, τα οποία δεν ε, μπορούν να βρουν τη συνένεσή μας και ούτε χωράει συμβιβασμό. Και δεν θέλει να κάνει βήματα προς την κατεύθυνσή μας στο Συμβούλιο. Το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ φιλόδοξο μέσα στο 2020 και πέρα από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη εγκρίνει, έχουμε πολλέ συναντήσει με εμπειρογνώμονε για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές. Περισσότερη δουλειά έχει ήδη γίνει. Τώρα πρέπει να πάρουμε τις σημαντικότερες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας συνοψίσατε το που βρισκόμαστε. Ε, δύσκολη κατάσταση. Να ακούσουμε τώρα και τους κοιόδες συζητητές για το ζήτημα από το ΕΛΚΟ. Κύριο Σαρθαλέχος έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την έκθεση, για τη δουλειά που κάνει στα πλαίσια του φακέλου δύσκολη δουλειά. Οι αρχικές θέσεις ε, απέκλειναν σημαντικά και αυτή η απόκληση εξακολουθεί να υφίσταται για μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε βεβαίως ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, σημαντική πρόοδος, και βεβαίως χρειάστηκε μακρά συζήτηση. Γι' αυτό όπως για το θέμα του ορισμού του όρου τρομοκρατία κρίσιμο ζήτημα για να μπορούμε να γνωρίζουμε τελικά ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Είναι δύσκολος επίσης ε, ο ορισμός της αρμόδιας αρχής για, τις, ε, για αυτή δηλαδή που θα εκδίδει τις ε, απόσυρσης περιεχομένου με το σχετικό περιεχόμενο Από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα της διασυνορικής συνεργασίας, άλλο δύσκολο ζήτημα. Ο κανονισμός αυτός ε, θεωρητικά θα πρέπει να επιφέρει προσθέμενη αξία στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και βεβαίως πρέπει να έχει μια διασυνοριακή διάσταση αυτές, οι διαταγές απόσταση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ε, εξετάζουμε διάφορους τρόπους για να συμβεί αυτό και οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ σίγουρα έχουν τη σημασία τους. Τώρα υπάρχει το θέμα των φίλτρων. Αφενό πρέπει να σεβαστούμε την αρχή σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ε, στους παρόχους υπηρεσιών μια γενική υποχρέωση παρακολούθησης ε, ελέγχου του περιεχομένου. Ε, από την άλλη θα πρέπει να γίνει και μια δουλειά σε επίπεδο πρόληψης όπως άλλωστε ισχύει και σήμερα. Θέλουμε λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση να περάσουμε από ένα σύστημα εθελοντικό στην πραγματικότητα σε ένα σύστημα που θα ρυθμίζεται καταλήλως Εμείς λοιπόν το ΕΛΚ θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη σημασία να βρεθεί μια λύση στο θέμα της διοσυνερικής ε, διάστασης αυτών των διαταγών απόσυρσης και να συνεχίσουμε βεβαίως να συζητούμε το θέμα των φίλτρων. Πιστεύουμε ότι και στα δύο αυτά σημεία ε, και για τα δύο αυτά σημεία υπάρχει περιθώριο ε, συμφωνίας με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να αναζητήσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Θαρθαλέχος για την ομάδα S&D, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Η κυρία Μαρίνα Καλιούραντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκη, τον εισηγητή, για την παρουσίασή του σήμερα, αλλά και για την όλη του στάση κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων στους τελευταίους 5-6 μήνες, ε, πώς ηγήθηκε αυτόν. Ε, ε, δεν συμφωνώ ότι έχει μπλοκαριστεί η, η όλη η υπόθεση. Αντιθέτως, έχει σημειωθεί πρόοδος, ε, έχουμε φτάσει σε συμβασμούς. Βεβαίως παραμένουν εκκρεμή ζητήματα που θα εξεταστούν στους τριμερείς διαλόγους. Βεβαίως, υπό την ηγεσία του κυρίου Γιάκη σημειώθηκε πρόοδος. Κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο για τρομοκρατικό περιεχόμενο διαδικτυακά. Πρέπει να αποσύρεται. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς αυτό το πολιτικό έγγραφο θα γίνει ένα έγγραφο που θα μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό, γρήγορο τρόπο που θα φέρνει αποτελέσματα. Και αυτό είναι το βασικό σημείο διαφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Κάποια από τα θέματα που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ε, να επιτρέψω την προσοχή όμως ε, και εγώ στο θέμα των διαταγών. Και εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ω ένα ενιαίος νομικό χώρο, Αλλά είμαστε ρεαλιστέ. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Είναι διαφορετικέ δικαιοδοσίε. Ε, δεν νομίζω λοιπόν να είναι αποτελεσματικό να εισαγάγουμε τώρα δεσμευτικά, δεσμευτικά διασυνοριακά μέτρα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν εδώ έχει μια σωστή θέση, κατά τη γνώμη μου, η οποία ε, εγκρίθηκε από, την προηγούμενη, το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Η εντολή μας είναι ισχυρή και βεβαίως στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να φτάσουμε σε συμβασμούς. Αυτοί οι συμβασμοί όμως δεν πρέπει να διακυβεύσουν το έργο ε, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι, πιο αποτελεσματικοί. Ε, ήταν πολύ ενθαρρυντικό το ότι ακούσαμε ότι η Επίτροπος Γιώχανσον προσωπικά ε, είναι πλάκη στην όλη διαδικασία. Αναμένω τη συνεργασία μαζί της. Θα έχουμε και μια νέα Προεδρία του Συμβουλίου και με αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι το παρόχρονο διάγραμμα με τον πρώτο τριμερή διάλογο τον Μάρτιο είναι σωστό Μα δίνει χρόνο να διαπραγματευτούμε και μεταξύ μα και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν για να βρούμε μια καλή συμβιβαστική πρόταση. Όπω είπα όμω, η ουσία είναι ότι δεν πρέπει εδώ να κρίνουμε απλά ένα πολιτικό κείμενο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η υποχρέωσή μα είναι να βρούμε λύσει, οι οποίε είναι αποτελεσματικέ, να είναι εφαρμόσιμε και που πραγματικά θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Διότι όλοι εδώ συμφωνούμε. Δεν υπάρχει περιθώριο για να για τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ και τώρα για την ομάδα Renew η κυρία Παγραθαρτουντούα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδελφούς. Συγχαίρω και εγώ τον κύριο Γιάκη. Εξαιρετική δουλειά. Και όλοι εμείς αισθανόμαστε ότι προσωπούμαστε ορθώς με όσα προωθεί. Πράγματι έχουμε σημειώσει πρόοδο και εγώ πιστεύω ότι το πνεύμα που μας κινεί όλους είναι να πετύχουμε να έχουμε βιώσιμες λύσεις. Λύσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν και αυτό που ανακρίνει το Κοινοβούλιο να μην είναι εμπόδιο, αλλά το αντίθετο. Εμείς ε, θέλουμε το τρομοκρατικό περιεχόμενο να εξαφανιστεί από το διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, είχαμε ένα έντονο χρονοδιάγραμμα και μπορούμε να πούμε ότι είναι ορθή, συνήθιση ταχύτητα που ακολουθείται και χάρη στο συμβασμό της Επιτρόπου Γιώχανσον, εγώ έχω ελπίδα ότι τους επόμενους μήνες, χωρίς να χάσουμε υπερβολικό χρόνο, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε θέματα που είναι πολύ πρόκειται να διαχειριστούμε τώρα λόγω των συγκρόμενων συμφερόντων ε, μεταξύ θέσης ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Εγώ ελπίζω ότι θα βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να επιλύσουμε τα δύο-τρία εκκρεμή ζητήματα που έχουμε στις διαπραγματεύσεις. Το βέβαιο είναι ότι αν μιλάμε για το διασυνοριακό καθεστώς, ε, ακόμη και όσοι είμαστε υπέρ πιο έντονης συνεργασίας, ε, βρίσκουμε ένα θέμα με τον ε, νομικό περιορισμό και θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο η παρέμβαση σε ένα δεύτερο κράτος από την πλευρά ενός κράτους ε, μέλους να υπάρξει να γίνει δυνατόν, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε αυτή τη δυνατότητα να συμβιβάσουμε τη μία και την άλλη θέση και γιατί είναι δυνατό αλλά και απαραίτητο γιατί θα πρέπει να τακτοποιήσουμε το διαδικτυακό χώρο και να αφαιρέσουμε το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Ευχαριστούμε τώρα για τους πρασίνους, ο κύριος Μπραΐερ. Ευχαριστώ. Τον εισηγητή, ο φάκελος αυτός αφορά το πώς θα συμφιλιώσουμε αποτελεσματικά την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και την προστασία των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Ε, και η ομάδα του Κοινοβουλίου διαπραγματεύεται βάσει μιας ε, θέσης που υθετήθηκε από αυτή την Επιτροπή και πολλοί από εσά που ήταν παρόντες υπερψήφισαν. Και ο στόχος της θέσης μας που διαφέρει όντως από την πρόταση είναι να διαφυλάξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα επιγραμμικά. Επομένως, έχουμε προτείνει αρκετές αλλαγές και στον ίδιο τον τίτλο του κανονισμού. Παραδείγματο χάρη, δεν θέλουμε υποχρεωτικά φίλτρα ανεβάσματος που θα οδηγήσουν σε μαζική εμπλοκή νόμιμου υλικού γιατί δεν θα μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο όπως μπορούν οι άνθρωποι και είναι πολύ εύκολο να καταστραγηθεί και μη αποτελεσματικό. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ε, που είναι κατά των φίλτρων και είναι απαράδεκτη η προσέγγιση αυτή. Θέλει επίση οι εντολέ αφαίρεση στο Κοινοβούλιο να εκδίδονται προεξάρτητα εκεί στη χώρα ε, όπου φιλοξενείται ε, στη χώρα κατοικίας του παρόχου και θέλουμε να έχουμε και ένδικα μέσα προσθέτει ένα προηγούμενο κανονισμό αυτό ε, για τη ρύθμιση παρανόμου περιεχομένου στο διαδίκτυο παγκοσμίω και γι' αυτό θέλουμε να το έχουμε σωστά. Οι χρήστε του διαδικτύου, οι επιχειρήσει, οι καλλιτέχνε και οι δημοσιογράφοι, οι ερευνητέ ε, και <clears throat> τα μέσα μαζική ενημέρωση μα παρακολουθούν. Έχουμε λάβει πάρα πολλέ επιστολέ και σχόλια και ε, γνωρίζουμε ε, τι θέλει η κοινωνία των πολιτών και ο κλάδος. Έχουμε λάβει επιστολές ε, και από τον Οργανισμό Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακόμη και τρεις ειδικοί ηγητές του ΙΕ μας ε, επενθύμησαν ότι είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τρομοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά πρέπει να προφυλάξουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς το Κοινοβουλίο θα πρέπει να σταθούμε ενωμένοι πίσω από τη θέση μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές επειδή το πράττουν αυτό και επειδή διαπραγματεύονται επί της θέσης αυτής. Εδώ διαπραγματευόμαστε περίπου για δύο μήνες και δεν έχει μπλοκαριστεί ο φάκελος αυτός σε καμία περίπτωση. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλά θέματα, όπως τόνισαν και οι συνάδελφοι. Στο τελευταίο τριμερή διάλογο είχαμε πραγματικό πνεύμα να βρούμε ένα κοινοτόπο, Καλά οδεύουμε με το φάκελο αυτό και εργαζόμαστε για πιθανούς συμβασμούς και εμείς στο Κοινοβούλιο. Το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου ως έχει θα έχει πολύ σημαντική προσθεμένη αξία ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Εμεί θα διασφαλίσουμε ότι θα αφαιρείται γρηγορότερα το τρομοκρατικό περιεχόμενο, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε ένα μηχανισμό αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσουμε το θέμα και στο εξωτερικό που δεν υπάρχει τώρα και θα θεσμικοποιήσουμε τη διασυνορική συνεργασία των αρμοδιών αρχών θα επιτρέψουμε οι αρχέ να επιβάλλουν μέτρα στου παρέχου για να αντιμετωπίσουν καλύτερα το δρομικροτικό περιεχόμενο επιγραμμικά. Παραδείγματο χάρη, οι χρήστε θα μπορούν ε, να στείλουν ένα μήνυμα ότι υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο και θα επιτρέψουμε καλύτερη δίωξη της τρομοκρατική υποχρεώνοντα υποχρεώνοντας ε, τα άτομα να καταγγέλουν το τρομοκρατικό περιεχόμενο και του παρόχου να καταγγέλουν το περιεχόμενο και παρέχοντα τα κατάλληλα δεδομένα. Εργαζόμαστε λοιπόν από κοινού να βρούμε λύσει που αποτελεσματικά θα αντιμετωπίσουν το δημοκρατικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι ακολουθούμε την ορθή εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Για το ID, ο κύριος Γκαρό, δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Να περάσουμε στην ΚΟΕ, στην κυρία Έρνστ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον εισηγητή, ο οποίος ήταν υποδειγματικός στον τρόπο με τον οποίο ηγείται σε αυτή την προσπάθεια. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Αυτό είναι ο δρόμος, πιστεύω, και έτσι θα προχωρήσουμε. Και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο αφήνει όλα τα εδεχόμενα ανοιχτά, όλους τους δρόμους, δεν κλείνει πόρτες. Θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά και να τον υποστηρίξω. Ένα αυτό. Δεύτερον, για μας είναι πολύ σημαντικό η κεντρική ιδέα της ε, άποψης του Κοινοβουλίου να διατηρηθεί. Ε, τα ακούσαμε ποια είναι αυτά. Δύο είναι τα σημαντικότερα που πρέπει να μείνουν στο κείμενο. Το πρώτο είναι βεβαίω θέλουμε να απομακρύνουμε τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο και δεν αμφισβητεί κανεί τίποτα, ούτε διαφωνεί στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διαφυλάξουμε και να σεβαστούμε την ανεξαρτησία των συστημάτων, ε, τις δικαιοδοσίες, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Ε, εκεί είναι η δυσκολία. Πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία. Γι' αυτό εξακολουθούμε να έχουμε επιφυλάξει σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές λύσεις. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να κάνουμε ε, κάποιες προσπάθειες για να βρεθεί ένα συμβιβασμό πάντα εφόσον διαφυλάσσεται αυτή η ισορροπία. Αυτό που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο είναι τα διάφορα φίλτρα για το τι θα ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Έχει λάβει θέση εδώ και ε, πολύ καιρό η διαδικτυακή κοινότητα. Και πραγματικά μένα, ακόμα με ενοχλεί και θυμώνω που πήραμε τόσο λάθος απόφαση για τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright. Δεν θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Αυτά τα φίλτρα είναι τελείως ακατάλληλα ως υποχρέωση. Το ξέρω ότι υπάρχουν τέτοια φίλτρα, αλλά να μην είναι υποχρεωτικά. Είναι ο πιο λαθασμένος δρόμος περιορίζεται και δυσκολεύεται η ελευθερία της έκφρασης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, της δημοσιογραφικής έκφρασης. Δεν είναι εδώ να έχουμε φίλτρα για το τι θα σηκώνει. Κατά τα άλλα ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα, δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε πολύ στη σημερινή ημέρη σε δέταξη. Έχουμε βαρύ πρόγραμμα Eurojust Μετά θα έρθει ο κύριος Δίδια Ρέντερ, ο Επίτροπος δικαιοσύνη και στη συνέχεια η Κροατική Προεδρία. Να προχωρήσουμε. Είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει τίποτα σύντομα. Η Επίτροπες Χάνσον μας είπε ότι είναι προθυμή να έρθει να φέρει επικοδομητικέ προτάσει για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην εντολή του Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο. Και μετά να ξανακούσουμε και τον εισηγητή μας. Ενθανητικά αυτά που ακούσαμε, παρά τις δυσκολίες που μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει. Ακούσαμε ότι οι συνάδελφοι εκτιμούν το έργο σας και είναι επικοδομητική η στάση. Πάρα πολύ σημαντικό για να γίνει σωστά η δουλειά. Σύντομα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην το πολύ καθυστερήσουμε. Δεν είστε και υποχρεωμένοι, αν θέλετε, αλλιώ δεν πειράζει. Ναι, να πω εν συντομία ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εξαιρετικό έργο της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον για το εξαιρετικό έργο του και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Υπάρχει εδώ βούληση στην αίθουσα για να φτάσουμε σε συμφωνία για αυτόν τον πολύ σημαντικό κανονισμό και αυτό είναι θετικό. Από την πλευρά μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος, όπως είπε και η Επίτροπός μας, Είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε την εξέβρεση εμβαστική λύση, να βρεθούν αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του τρομοκρατικού περιεχομένου επιγραμμικά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σύντομοι. Κύριε Γιάκη, θέλετε το λόγο. Βλέπω ότι και κάποιος ε, σκιώδης συγητής εδώ ε, προσέγγισε το ζήτημα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσω στα πολωνικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους για την επικοδομητική τους στάση. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος ε, για το πώς συνεργάστηκε η ομάδα σε αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί υπάρχει βούληση να φτάσουμε σε συμβασμούς. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να ληφθούν σημαντικότατες αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον της ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αυτά τα δύο θέματα που εκκρεμούν ε, είναι πρωτοφανή. Μέχρι τώρα δεν έχουν συζητηθεί, όπως ε, παίρνουν χάρη, η διασυνοριακή εντολή αφαίρεσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Χρειαζόμαστε ευρία πλειοψηφία για την απόφαση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο για αυτά τα δύο εκκρεμή ζητήματα και το Συμβούλιο γνωρίζει ότι σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο πρόκειται για θέματα πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο και εμεί θα εργαστούμε για το συμβιβασμό. Ακούσαμε πώς έχει η κατάσταση και όπως είπα θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάκη για το συμπέρασμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο 8, αποστολή της Επιτροπής Λίμπε στη Γιουρούτζα, στις Χάγη, στις κάτω χώρες, που έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου. Έχουν παρουσίαση του σχεδίου απολογισμού της αποστολής. Πρόκειται για μια κοινή συζήτηση με το σημείο 9, ανταλλαγή απόψεων με τον προσκεκλημένο μα σήμερα τον κύριο Λάντισλαβ ε, Χάμραν, που είναι πρόεδρος της Eurojust. We welcome Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της ε, Eurojust, ε, σημαντικό οργανισμό στο σύνολο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το έργο σας για τη δική μας επιτροπή. Καλώς ήρθατε κύριε Χάμραν. Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του νέου κανονισμού της Eurojust 2018 που άρχισε να εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο του 2017, Συγγνώμη. Έχουμε καλή ευκαιρία ο πρόεδρος της Eurojust να μας ενημερώσει για την κατάσταση της εφαρμογής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της θέσης της Δανίας στη Eurojust έχει λάβει χώρα ε, λόγω της λησφωνοποίησης, λησαβωνοποίησης. Επίσης, είναι καλή ευκαιρία να μας μιλήσετε για τη συνεργασία της Eurojust με τις τρίτες ε, χώρες, καθώς και στο παρελθόν έχουμε συζητήσει για πολλές συμφωνίες Eurojust με τρίτες χώρες, όπως η Ελβανία, η Γεωργία και η Σερβία. Λοιπόν, καταρχήν, να ακούσουμε σχετικά με την έκθεση της αποστολής, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παζ Γασαρτούντου, που ήταν επικεφαλή αυτής τη αντιπροσωπείας και στον κύριο Βίντσε και κατόπιν ε, θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Eurogist και θα έχουμε μια συζήτηση ε, μέχρι τις 10 ε, και 4 όταν θα έρθει ο Επίτροπος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να πω ότι η αποστολή μας έλαβε χώρα με κανονικότητα. Ένα γενικό ζήτημα είναι το εξής. Είχαμε μια καλή εντύπωση τους ατζέντα εργασία ήταν πλήρης με πολύ συγκεκριμένα σημεία και η εντύπωσή μας σε σχέση με τη Διευθυντική Επιτροπή της Eurojust ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ δυναμική η ομάδα, ιδιαίτερα ε, προδραστική, ότι αναζητά τις καλύτερες ε, ευκαιρίες για το τι μπορεί να κάνει η Eurojust, ε, αν λάβουμε υπόψη ότι έχει και σημαντικό άχθος εργασίας, σε ένα πλαίσιο που το οργανωμένο έγκλημα συγκεκριμένα έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο πολύπλοκο ως προς την προσέγγισή του. Και επομένως οι προσπάθειες της Eurojust και οι πραγματικές υποθέσεις ε, επί των οποίων εργάζεται η Eurojust είναι πιο, πιο πολύπλοκες. Μας ε, έδωσαν παραδείγματα συγκεκριμένων υποθέσεων, μπορούσαμε να δούμε ε, πραγματικές προσωμιώσεις. Όλα αυτά ήταν πολύ ικανοποιητικά για κάποιες πολύ πολύπλοκες μορφές εγκλημάτων και επίσης ε, μας μίλησαν και για τις πραγματικές ανάγκες σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε επίπεδο πόρων, πληροφορικής, σε επίπεδο πραγματικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι οργανισμοί που είναι σημαντικοί για το θέμα της ασφάλειας και για τη δικαστική αστυνομική συνεργασία, θα έβλεπαν αύξηση στον προϋπολογισμό τους. βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανομαλία εδώ στην περίπτωση της Eurojust. Αυτό μας το εξέφρασαν ε, ανοιχτά και ειλικρινά και φαντάζομαι ότι σήμερα θα συζητήσουμε κάποια στιγμή και αυτό το θέμα. Εμείς μείναμε πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που συζητήσαμε ε, το θέμα της, ε, του θεματολογίου και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η Eurojust. Επίσης, θέλουμε να διαβάσουμε στους συναδέλφους ότι μιλάμε για τα θεμελιώδη ζητήματα της δικαστικής συνεργασίας όπως το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας ή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που σίγουρα είναι ένας σημαντικός μηχανισμός ε, συνεργασίας Όμως ε, έχοντας κατά νου αυτές τις νέες μορφές εγκλήματος και πώς έχει μεταμορφωθεί η κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια, πράγματι η Eurojust ε, κάθε φορά έχει όλο ένα και μεγαλύτερο άχθος εργασίας. Επομένω, μα είπαν ότι του τελευταίου 6 μήνες έχουν λάβει πάνω από 900 υποθέσει ε, ευρωπαϊκού εντάλματο σύλληψη. Επίση, ε, συζητήσαμε αυτό το θέμα τη αμοιβή εμπιστοσύνη που βρίσκεται στη βάση αυτού του μηχανισμού. Και μιλήσαμε για την αναγκαιότητα των γενικών εναρμονήσεων. Κάτι που το βλέπουμε σε όλα όσα αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και το διεθνές έγκλημα. Επίσης, ε, να πω κάτι σημαντικό για το θέμα Πρόκειται για το να μην μπούμε σε κανένα είδους διένεξης ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καθώς η φιλοσοφία με την οποία ξεκινά δεν είναι ακριβώς ίδια με τη Eurojust. Η Eurojust βασίζεται στα εθνικά κράτη, δεν έχει όμως πόνδια όραμα. Για τα οικονομικά ζητήματα νομίζω ότι θα συζητηθούν ε, αυτά τα θέματα από τους συναδέλφου. Όπως σας είπα, ήταν εξαιρετική η εντύπωσή μας για το χειρισμό των υποθέσεων και ευχαριστούμε επειδή μας δώσατε ένα μια πραγματική παρουσίαση για το πώς είναι ε, ο χώρος ε, και για το θέμα του εγκλήματος και επίσης ε, πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη και να μην υπάρχει ατιμορρησία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δικαστική συνεργασία και τον μέσων που έχουμε όπως το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, ή το πώς θα γίνει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συναγγελία. Είναι θέματα που μας αφορούν και τα εξετάζουμε στη σχέση μας. Αλλά πολύ συγκεκριμένα θέματα τεχνικής ε, φύσεως ε, είναι τα εξής. Όλα όσα έχουν να κάνουμε τα συστήματα τα ψηφιακά συστήματα, τα διαδικτυακά συστήματα, όλα όσα χρειάζονται επικαιροποίηση. Αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούμε να χειριστούμε ε, το μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Χρειάζονται και οι κατάλληλοι πόροι για την επικαιροποίησή τους. Έχουμε φυσικά και το θέμα της ψηφιακής ε, ποινική δικαιοσύνη. Για όλα αυτά χρειάζονται τεχνικές ε, τεχνική πρόοδος, γιατί διαφορετικά στο μέλλον μπορεί να μείνει αναποτελεσματική η Eurojust. Όλα αυτά μας παρουσιάστηκαν. Αυτή είναι η σύνοψή μου. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Βίντς επίσης ήταν μέλος της αντιπροσωπείας αυτής. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες πτυχές τη αποστολή μα ε, θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ ήταν μια πολύ καλή αποστολή με τη συνάδελφο να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χάμπραν και την ομάδα τη Eurojust που μας έδωσαν μια συνολική ε, και χρήσιμη εικόνα των δραστηριοτήτων της Eurojust ε, εντυπωσιαστήκαμε διότι είναι πολλές και ποικίλε οι υποθέσεις 6.500 μόλις ε, το 2018 είναι εντυπωσιακό για μια υπηρεσία με 300 άτομα προσωπικό. Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των εσωτερικών δομών Eurojust το γεγονός επίσης ότι ουσιαστικά είναι ένα απόθεμα γνώσεων ε, με τις υποθέσεις αυτές που μπορεί να μοιραστούν με τα κράτη-μέλη. Ε, για να αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Eurojust και άλλων ε, υπηρεσιών στον τομέα τη δικαιοσύνη των ιστορικών υποθέσεων. Πρόκειται για παίκτε κλειδιά στην ίδια αλυσίδα ασφάλειας και βεβαίω στην πρώτη γραμμή είναι η Eurojust, στην τελευταία γραμμή μάλλον, είναι εκεί που μπαίνει τέλο υποθέσεις υποθέσει αυτέ με την δίωξη ε, είναι πολύ στενή συνεργασία με την Europol και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα στον τομέα του εγκλήματος, της τρομοκρατίας, ε, πνευματικής διοκτησίας κλπ. Ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λυπούμεθα που δεν είναι στην ίδια πόλη αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο θεσμοί, ε, μιας και ουσιαστικά κινούνται στο, στο ίδιο πεδίο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ε, παρά την απόσταση που υπάρχει τη γεωγραφική. Επίσης ε, υπάρχει και μια κάποια επικάλυψη μεταξύ των δύο αυτών ε, οργάνων. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό όταν θα αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα έχουμε και τις αιτήσιε εκθέσεις και από τις δύο υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά την εξοδαφική συνεργασία, μια σειρά από συμφωνίες με τρίτες χώρες έχουν συναυθεί. Ε, παραδείγματα ε, εξαιρετική συνεργασία με τρίτε χώρε. Δεν σταματάει το έγκλημα στα σύνορά μα, ούτε στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Προσπαθεί λοιπόν η Eurojust να επεκτείνει το διεθνές δίκτυο συνεργασίας ε, με τρίτες χώρες, κρίσιμη, αυτέ αυτές τις συμφωνίες συνεργασίες, μιας και έχουμε όλο και περισσότερες υποθέσεις που αφορούν τρίτες χώρες. Το 2018 είχαμε μια σημαντική αύξηση. Ενθαρρύνουμε την Eurojust ε, να έχει μια καλύτερη πολιτική επικοινωνίας διότι μετά από κάποιες σημαντικές υποθέσεις τα κράτη-μέλη είναι αυτά ε, τα οποία ρέπουν τις δάφνες των επιτυχιών. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ε, ότι συμμετείχε ε, και συνεισέφερε με καθοριστικό τρόπο ε, η Eurojust με την δικαστική συνεργασία που πρόθεσε. Χρειάζεται λοιπόν επικοινωνία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η Eurojust μας είπε ότι θα μπορούσε να μας παρουσιάσει κάποιες σημαντικές υποθέσεις ενδεχομένως και κλεισμένων των θυρών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Τώρα το θέμα το δημοσιονομικό επίσης πολύ σημαντικό. Η Eurojust είναι ένα μικρό μέρος του προπολογισμού της αλυσίδας της ασφάλειας ε, είναι πολύ μεγάλο φόρτο εργασία και αυτή η αύξηση μόλι 1% του προπολογισμού Eurojust ε, για το, στα πλαίσια του επόμενου, του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, ενώ έχουμε αύξηση των, της νομολογίας σε διψήφιους αριθμούς, θα δυσκολέψουν όλα αυτά το έργο της Eurojust. Προκύπτουν και νέες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια, ε, τρομοκρατία, κυβερνοέγκλημα, ε, εμπορία μεταναστών. Ε, θα είναι λοιπόν καλό να δούμε, να μας πει ο κ. Χάρμαν πώς βλέπει το θέμα της χρηματοδότησης πιο μακροπρόθεσμα, διότι υπάρχουν και προτάσεις στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα συνεχίζουμε, θα συνεχίσει η ομάδα μας να είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο από την αποστολή, από τα μέλη της αποστολής ε, στην Χάγη ε, να ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον πρόεδρο της Eurojust. Ε, καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξή σας στον προπολογισμό του 2020 και πρέπει να πω ότι χάρη στη δική σας υποστήριξη έχουμε μια πολύ καλύτερη, έχουμε πολύ καλύτερες δημοσιονομικές προοπτικές για αυτό το έτος. Θέλω να ευχαριστήσω και την, την Μάιτε και τον Λοράν για τις πολύ καλές συζητήσεις που είχαμε. Μάθαμε πολλά από εσά και ελπίζουμε και εσείς κάτι να μάθατε από μας. Όλα όσα ελέγχθησαν ε, τα επιβεβαιώνω. Επίσης ε, ισχύει ε, αυτή η η προσφορά μας να έρθουμε στην Λίμπε για να σας μιλήσουμε για κάποιες σημαντικές υποθέσεις με τις οποίες ασχολούμαστε, εφόσον το επιθυμείτε. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση της αποστολής σας, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Θα ήθελα όμως ε, σήμερα να δώσω εγώ μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα αυτά. Θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν ήταν ποτέ τόσο καλή όσο σήμερα και τόσο έντονη. Τα στοιχεία ε, μπορείτε να δείτε ότι το επιβεβαιώνουν. Ε, τα κράτη-μέλη συνεργάζονται όλο και περισσότερο και αν δούμε τι συνέβαινε πριν από 20 χρόνια, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκό Έντελμα Έρευνας, δεν υπήρχε Eurojust, ε, δεν υπήρχαν κοινέ ομάδε έρευνα. Κατά τη γνώμη μου, πραγματικά πάμε προς σωστή κατεύθυνση. Πάμε από την απομόνωση στη συνεργασία. Βεβαίως έχουμε προκλήσεις μπροστά μας, αλλά υπάρχουν και επιτεύγματα. Υπάρχουν και επιτυχίες και αυτό χάρη και στην δική σας υποστήριξη και τη δουλειά σας. Σε ό,τι αφορά δύο υποθέσεις ε, ε, που ξεκίνησαν πέρυσι από τη Eurojust, ε, είχαμε 4.000 μάλλον νέες, θέσεις, υποθέσεις, συγγνώμη, και μαζί με αυτές που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα έχουμε φτάσει στις 8.000. Οι περισσότερες προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά έχουμε και από τρίτες χώρες υποθέσεις. Ε, υποστηριζουμε υποστηρίζουμε ένα κράτη-μέλη ε, σε 1.400 περίπου επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας. Οργανώσαμε 430 συνεδριάσεις ε, συντονισμού. Εκεί ε, οι εισαγγελεί, οι ανακριτές, ε, οι ερευνητέ αντέλεξαν πληροφορίες ε, για διάφορες πτυχές του, της υπόθεσης. Έπρεπε να μιλήσουμε μεταξύ του, διότι υπήρχαν παράλληλες έρευνε, Έπρεπε να επιλύσουμε και κάποια ζητήματα ε, σύγκρουση δικαιοδοξιών για το υπήρχε ένα θέμα δηλαδή του ποιο ηγείται ε, κάποιων εγκληματικών οργανώσεων. Υπάρχουν και διαφορέ στα νομικά συστήματα συζητήσαμε τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ε, πότε να χτυπήσουμε ε, την ε, οργανωμένη αυτή, τις οργανωμένες αυτές εγκληματικές ομάδες, πότε να προβούμε σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, πραγματικά είναι νομίζω αρκετά εντυπωσιακά αυτά. Αποτελέσματα των κρατών μελών, εμείς απλώς βοηθούμε τα κρατημέλη να πετύχουν τους στόχους αυτούς. Ε, σε οκτώ υποθέσεις ε, συμφωνήσαμε πότε θα ε, διώξουμε έναν ύποπτο. Συλλάβαμε πάνω από 2.500 υπόπτους και διευκολύναμε χιλιάδες ευρωπαϊκά ατλήματα σύλληψης, ευρωπαϊκά ατλήματα έρευνας, ε, και αιτήματα αμοιβαία ε, δικαστική συνδρομή. Θέλω θα να αναφερθώ πραγματικά στη σημασία των κοινών ερευνητικών ομάδων, διότι αυτέ οι ομάδε παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση του συνοριακού εγκλήματο. 272 κοινέ ομάδε έρευνα υποστηρίχθηκαν από τον κύριο Τζάστο, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο, σε επίπεδο πραγματογνωμοσύνης Κατά τη γνώμη μου αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η έννοια της δικαστικής συνεργασίας λειτουργεί και στην πράξη. Και αυτά που μπορεί να πετύχουν τα κράτη-μέλη ε, με τη βοήθεια μέσα υπηρεσίας προς Eurojust ε, τα βλέπουμε μπροστά μας. Είναι σημαντικό επίσης ε, και λέω ξανά και ξανά ότι είναι τρεις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το θέμα είναι, το πρώτο, το ένα είναι η παγκοσμιοποίηση, διότι σύνορα υπάρχουν όλο και λιγότερο, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την ανάγκη αυτών των στοιχείων, ε, ψηφιοποίηση, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας, ε, ιδιαίτερα όταν πρέπει να ανταλλάξουμε ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, αυτό αφορά πολλά γιγαμπάιτ και τεραμπάιτ δεν υπάρχουν ασφαλή διάβλη επικοινωνία ε, για να, που να μπορούν να υποστηρίξουν την ανταλλαγή τέτοιου είδου φακέλων σε τέτοια κλίμακα. Έχουμε ξεκινήσει και ένα σχέδιο ψηφιακής ποινική δικαιοσύνης ε, για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και το τρίτο βέβαια και εξαιρετικά σημαντικό επίσης για κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης είναι το θέμα των πόρων, των οικονομικών πόρων μεταξύ άλλων ε, εμείς θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Κάναμε τη δουλειά μας. Μεταρρυθμίσαμε την οργάνωσή μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, για να μπορέσουμε να διαθέσουμε ακόμα περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο φόρτο εργασία. Σα ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Αναμένω τα ερωτήματά σα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή τη Eurojust. Το μόνο που εύχομαι είναι εμείς οι ευρωβουλευτές να προβάλλουμε περισσότερο το έργο τους Eurojust, ε, να ενημερώνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί δικαιούνται να γνωρίζουν ε, το μέγεθος της πρόκλησης και πώς μπορεί να αποκριθεί ε, η Eurojust τι κάνει, πώς ε, προχωρεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέχρι και συλλήψεις. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο συζητούμε. Και εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό. Αλλά εκείνοι καθημερινά κάνουν αυτή τη δουλειά. Τώρα έχει έρθει η ώρα των μελών της Επιτροπής μας να σχολιάσουν. Επιμένω ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και είναι δικό μας καθήκον να τους ενημερώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Τι υπάρχει, τι λειτουργεί, τι δουλεύει, τι κάνει η Eurojust. Η δουλειά μας είναι. Ποιο θέλει το λόγο, παρακαλώ. Για να σχολιάσετε αυτό που ακούσαμε το σχέδιο έκθεσης και ε, την αναφορά της αποστολής στη Χάγη. Ο κύριος Κρίς Πέτερς, παρακαλώ. Uh, Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της Eurojust. Όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το όργανο αυτό και θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο περισσότερο για αυτή τη φανταστική δουλειά που κάνετε πολλά χρόνια τώρα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε κι εσείς στη χρήση ηλεκτρονικών ε, δεδομένων ως ε, αποδεικτικών στοιχείο. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Ότι ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια δεδομένα όταν δεν απαγορεύεται, αλλά κάποια άλλα δεν μπορείτε γιατί απαγορεύεται. Πώς βρίσκεται η κατάσταση και πώς έχει. Ένα δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ε, πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας όπως την κάνατε στο παρελθόν, χρειάζονται απαραίτητοι οικονομικοί πόροι. Και θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στον προπολογισμό του Frontex, που είναι αρκετά Υψηλό και τον προπολογισμό για σας. Ε, ποια είναι η άποψή σα σχετικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Χαίρομαι που ακούω ότι η χρήση της Eurojust και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δεκτικών αρχών αυξάνεται. Δηλαδή όλο και περισσότερο καταφεύγουν σε εσά. Ακούμε όμως ότι δεν υπάρχει συνεργασία ή υπολείποτε γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουν ε, ε, επιτόπου στα κράτη-μέλη αρμόδιοι την ύπαρξη καν ε, των ε, διαφόρων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Πώς πρέπει να καταρτήσουμε και να εκπαιδεύουμε καλύτερα το προσωπικό στα κράτη-μέλη για να ξέρει ε, τι μέσα έχει και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Ποιες μορφές υπάρχουν δηλαδή στη δικαστική συνεργασία. Επίσης θα ήθελα να επανέλθω σε ένα από τα τελευταία που είπατε στην παρουσίασή σας όπου ε, κάνατε λόγο για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και τον όγκο των δεδομένων που πολλές φορές σας κατακλείζει. Καμιά φορά γιατί δεν υπάρχουν και ασφαλείς διαβλή διαβίβασης των δεδομένων. Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή στα κράτη-μέλη, στη Europol, στην ανταλλαγή και πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος ε, Τιντοράτση. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της Eurojust για το έργο σας. ακολουθήσω την πεπατημένη των συναδέλφων. Ξέρετε ότι και εμεί εδώ συζητάμε για το θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων ε, και για την ε, νομοθεσία για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Πριν έρθετε, ακριβώς ε, είχαμε τέτοιες ε, συζητήσεις ε, για το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για το ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα διασυνορικά εργαλεία που σας λείπουν ε, που πιστεύετε ότι θα χρειάζονται να εισαγγελείς, οι ανακριτές για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται για τις έρευνες σε ποινικές υποθέσεις και πώς εσείς βλέπετε να εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις σε αυτούς τους δύο φακέλους και πάλι από επιχειρησιακή σκοπιά, πιστεύετε ότι υπηρετούμε τις ε, ανάγκες που έχετε για θέματα ερευνητικά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Κινίτση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Χαμράν ε, για την παρουσία του εδώ και για τη σημαντική συνεισφορά της Eurojust στη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Χαίρομαι που μας είπατε ότι συνεχίζεται η συνεργασία αυτή και βελτιώνεται. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Παχαζαρτουντούα για την ε, σύνοψη και τους ε, συναδέλφους ε, που συμμετείχαν στην αποστολή. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον Διευθυντή. Καταρχήν, πάντοτε έχοντας κατά νου να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, ε, που είναι τόσο ε, σοβαρό θεωρείται ότι γενικά σήμερα χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία νομοθεσία που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με έναν πιο ομοιόμορφο τρόπο, δηλαδή μία πραγματική στρατηγική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης, Έχω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση σε ό,τι αφορά ε, τα καθήκοντα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Εσείς υπογραμμίσατε ε, την δυσκολία που μπορεί να συναντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Και φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σχετικό ζήτημα, όχι μόνο για τα ε, οικονομικά εγκλήματα, αλλά και άλλα εγκλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα και την τρομοκρατία. Εσείς, ε, βάσει της εμπειρίας της Eurojust, θεωρείτε ότι υπάρχουν σημεία ε, με άλλες 50 ε, χώρες και πώς θεωρείτε ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Καφιέρα Τεράου, ο επικεφαλής της Αγγελίας κατά της μαφίας, αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει στην Ιταλία, δηλαδή στον φιγούρα του συντονιστή δικαστή που συντονίζει τονίζει την δράση κατά της μαφίας ε, μεταξύ Ιταλικών και Νιγηριανών αρχών. Πιστεύετε ότι χρειάζεται ένας τέτοιος θεσμός για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες συντονισμού κατά πολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος με τις τρίτες χώρες. Επίσης, ε, να πω ότι συμφωνώ όσο υπόθηκαν από τη συνάδελφο Παχασαρτουντούα και με όσα είπατε εσείς ε, σε σχέση με τη συνεισφορά της Eurojust ε, να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες σας ε, και πρέπει να έχετε τους απαραίτητους πόρους και σίγουρα θα έχετε την υποστηρίξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριο Σαρσαλέχος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα την ε, έκθεση που εκπώνησαν οι συνάδελφοι και επίσης είναι πολύ ικανοποιητικό να ακούμε τα λόγια του Διευθυντή της Eurojust για την κατάσταση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έχει μόνο μία απάντηση που είναι να προωθήσουμε, διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τις ε, διαδικασίες συνοριακή συνεργασία. Υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι η Eurojust είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν χρησιμοποιείται αρκετά. Λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά της, όπως αντικατοπτρίζεται τα δεδομένα, θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε η Eurojust να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό της προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία που εν τέλει έγκυται στην εμπιστοσύνη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις προκλήσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος της Eurojust για το μέλλον. Μας αφορούν και μας ε, λόγω του νομικού θεματολογίου που πρέπει να αναπτύξουμε και φυσικά συνδέονται στενά με την ε, παγκοσμιοποίηση της ψηφιοποίηση και την ψηφιοποίηση. Εν ώψη λοιπόν αυτών των προκλήσεων θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη του πρέδρου της Eurojust σχετικά με τις δυσκολίες που ενέχει η έλλειψη εναρμόνισης τόσο στον ποινικό τομέα όσο και στον ε, δικονομικό τομέα μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών ε, νομοθεσιών. Και ε, θα θέλαμε να μας πείτε πού πρέπει να προωθήσουμε τη διαδικασία εναρμόνισης σε αυτούς τους τομείς. Κύριε Ρατσιβάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφθηκα την Eurojust και ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Συμφωνώ πολύ με το μήνυμα του Προέδρου ότι εμείς θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και να γίνεται γνωστή η ύπαρξη και το έργο της Eurozone. Ο κύριος Χάμρατ να αναφέρθηκε σε τρεις προκλήσεις και ξέρω ότι είναι πάντα δύσκολο για ένα οργανισμό ευρωπαϊκό να μιλάει για πόρους, είτε αυτή είναι ανθρώπινη είτε οικονομική. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ρωτήσω εγώ γι' αυτό και να μας δώσετε περισσότερες ε, πληροφορίες. Και όταν εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε το διασυνοριακό έγκλημα, θέλουμε να σας βοηθήσουμε και να είναι η προσπάθεια αυτή βιώσιμη και στο μέλλον. Και να μην έρχεστε συνέχεια να ζητάτε περισσότερα. Αυξήθηκε ο προπολογισμό της ε, ε, Ευρωπόλ και θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέλλον. Θα ήθελα παρακαλώ να μας πείτε ε, κάτι σχετικά. Η κυρία Ενετφέλτ είδα και το δικό σας χέρι. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Χάρμαν για την παρουσίαση. Ένα σχόλιο και ένα ερώτημα. Σας να πω, έχω αυτό που είπαν και άλλοι συναδελφοί για τα μέσα που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας. Εμείς σας υποστηρίζουμε. Αν μπορείτε να μας πείτε όμως και κάτι περισσότερο για το μηχανισμό το δημοσιονομικό, διότι αν κατάλαβα καλά η Eurojust ε, βρίσκεται σε μια ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή και αυτό δεν βοηθάει πολύ. Κάτι άλλο τώρα μπορείτε να μας πείτε για τις εξελίξεις σε κάποια κράτη-μέλη όπου οι κυβερνήσεις ε, όλο και περισσότερο ελέγχουν ε, και το δικαστικό τομέα και τις εισαγγελίε ε, ειδικότερα. Έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού. Μάλιστα, δεν λέω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Κύριε Χάμντρα, αν είδατε ότι υπάρχει υποστήριξη. Αν θέλετε το λόγο, ναι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο νωρίτερα, αλλά δεν με είδατε μάλλον. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την παρουσίαση και για το έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε τα καλά νέα, να, μαθαίν, να μαθεύονται τα καλά νέα και χρειάζεται βεβαίω περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία και ισχυρότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι δουλειά όχι μόνο δική μα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ε, και καθήκον ε, των αρμόδιων αρχών στα κράτη-μέλη. Η Eurojust λοιπόν χρειάζεται να έχει ισχυρή φωνή και στα κράτη-μέλη. Ήθελα να θέσω κάποια ζητήματα. Ε, Πρώτον, τον Δεκέμβριο στη Eurojust έλαβε χώρα μια μετάβαση ε, προς μια μόνιμη, προς ένα μόνιμο θεσμικό όργανο στη Χάγη ε, με εκπροσώπους των κρατών μελών. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτή τη μετάβαση, πώς αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο εργασίας σας, έχετε ε, διαπιστώσει ότι λαμβάνουν χώρα αλλαγές και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς για την Europol παραδείγματο χάρη έχετε κάποιο σχόλιο και κάτι ακόμα για το δημοσιονομικό πώς βλέπετε την κατανομή εργασιών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν κύριε Χάμπτραν όπως βλέπετε κάθε φορά ε, που υπάρχει έκθεση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ για το θέμα το δικό σας ε, ανανεώνουμε την υποστήριξη στον οργανισμό σας ε, όμως 10 ε, και 4 προβλέπετε η συζήτηση με τον Επίτροπο Reinders ε, που είναι ήδη εδώ, καλώς ήρθατε έχετε λοιπόν 10 λεπτά για να απαντήσετε όσο καλύτερα μπορείτε στα ερωτήματα που τέθηκαν για τα αρμοδιότητες της Eurojust έχετε το λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ για όλα τα ερωτήματα όταν πρέπει να απαντήσω μπροστά στον επίτροπό μου, έτσι είμαι κάπως πιο νευρικός. Ε, λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με το ερώτημα του κυρίου Πίτερς ε, ε για, το, για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων για όσους δεν γνωρίζουν αυτές τις δύο έννοιες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ό,τι αφορά το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων σε, υπάρχει μια ομάδα χωρών όπου μόνο ό,τι προβλέπει ο νόμος θεωρείται παραδεκτό αποδεκτικό στοιχείο. Ε, ό,τι δεν αναφέρεται στον νόμο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ε, μετά όμως έχουμε μια άλλη ομάδα χωρών, οι σκανδιναβικές χώρες, παραδείγματος χάρη, όπου οτιδήποτε είναι παραδεκτό εφόσον δεν απαγορεύεται από τον νόμο πρέπει να πω ότι από αυτού προκύπτουν ευκαιριακά κάποια ζητήματα ε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ε, ο διάλογος μεταξύ δικαστικών αρχών, μεταξύ εισαγγελέων ε, διότι όλες αυτές οι διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν με αμοιβαία κατανόηση, με διάλογο. Αυτό είναι και ο ρόλος της Eurojust, των συνεδριάσεων συντονισμού αυτών. Δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει το ζήτημα αυτό και βεβαίως εμείς είμαστε ρυθυμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας επ' αυτού. Για τον προϋπολογισμό τώρα και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά χαμηλό για μας ανησυχούμε διότι αυξάνεται ο φόρτος εργασίας, ο αριθμός των υποθέσεων αυξάνει κάθε χρόνο ε, και η αύξηση, η αύξηση αυτή είναι διψήφια. 17% πέρυσι και πρόπερσι. Δυστυχώς οι δημοσιονομικές αρχές ε, δεν ε, δεν σκοπεύουν να μας δώσουν περισσότερα χρήματα, όμως ο διάλογος με την Κομισιόν, με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο εδώ είναι κρίσιμος. Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που κάνουμε και γιατί είναι σημαντικό να εξισορροπήσουμε το πολιτεύσιο πλαίσιο, τα μέσα που διατίθενται, να δοθεί έμφαση στη δικαστική συνεργασία, όχι μόνο ε, στη συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου. Η κυρία Ζίπελ ρώτησε για την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Ε, η καλύτερη συγγνώμη κυρία Σίπελ σας απαντάει απαντάει στο ερώτημά σας ο κ. Χάμπτερ ναι συγγνώμη δεν είχα δει ότι μιλούσατε και εγώ απαντούσα με τη σειρά ε, λοιπόν χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση η καλύτερη προώθηση ε, της προσταμένης αξίας μας, η απόδειξη της προσταμένης αξίας είναι όταν ε, μπορούμε να βοηθήσουμε τους αξιωματικούς ε, των διαφορών κρατών μελών και μπορούν να το δουν αυτό. Πρέπει να γνωρίζουν όμως ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ε, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Europol, Eurojust. Οπότε πάντα ζητώ περισσότερα χρήματα για την CIPOL ή την EGTN, διότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις, τους ασφαλείς, ε, τους διάβολους επικοινωνίας, ε, ξέρετε ότι υπάρχει ένα δίκτυο ε, για τις αρχές που του νόμου. δεν υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο Eurojust, σε επίπεδο δικαστικών αρχών. Θα θέλαμε ακριβώς το ίδιο. Να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουν, την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία, τις τεχνικές λύσεις που έχουμε διαθεσή μας, ακόμα ε, και το CNN δεν μπορεί ε, να, ε, να ελέγξει, να επεξεργαστεί μεταφορά φακέλων μεγάλων μεγάλων μεγάλων μεγέθους οπότε αυτό το θέμα θα το βρούμε μπροστά μας τώρα τι λείπει ποια είναι τα εργαλεία που μας λείπουν τα τελευταία δέκα χρόνια Νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει ένα πολύ καλό πακέτο νομικών μέσων και αυτό το πακέτο είναι αρκετά πλήρες. Ε, δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα σε κάποιο μέσο, σε κάποιο εργαλείο το οποίο να μας λείπει. Ίσα ίσα νομίζω έχουμε, ότι έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που το σημαντικό είναι να ενδυναμώσουμε ε, αυτά τα μέσα και να τα απλοποιήσουμε. Ε, και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαφορών νομοθετημάτων στα κράτη-μέλη θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά αυτά τα ευρωπαϊκά ε, νομικά μέσα και πρέπει και αυτό να αποτελέσει προτεραιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες ε, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολύ καλό το ερώτημά σας. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια, ε, στην νομική μου είχαν πει ότι υπάρχουν δύο θέματα στο διεθνές δίκαιο. Ε, ε, τα κράτη και οι διεθνείς οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αποτελεί μέρος καμιά σύμβαση δικαστικής συνεργασίας. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει μια δουλειά σχετική, έχουν υποβληθεί προτάσεις για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μία από τις προτάσεις είναι τα κράτη-μέλη να αναφέρουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως αρμόδια εθνική αρχή ε, για την ε, αντιμετώπιση εγκλημάτων ΦΠΑ για πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Το θέμα είναι πώ θα, πώς θα αντιδράσουν τρίτες χώρες. Εμεί μπορούμε να τη δηλώσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το θέμα είναι θα το δεχτούν οι τρίτες χώρες. Αυτό θα το δείξει ο χρόνο. Ε, είναι και ένα θέμα που μα ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει πώ οι τρίτες χώρε θα αντιδράσουν σε αυτήν την έτσι ε, κάπως ασυνήθιστη έννοια, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο ομοσπονδιακό μοντέλο, αλλά δεν είναι ομοσπονδιακή ε, η δομή της Ένωσης. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα, σε σχέση με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και, αλλά και με τα κράτη-μέλη, αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη να έχουμε ε, αποδεικτικά στοιχεία, να εκτελέσουμε κάποια εντολή, κάποιο ένταλμα σύλληψη με τρίτη χώρα. Οπότε πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Να μην έχουμε μόνο ε, σημεία επαφή σε 52 τρίτε χώρε, να έχουμε περισσότερε συμφωνίε συνεργασία με τι τρίτε χώρε αυτέ. Ε, συνεργασία που να μην είναι μόνο ad hoc, να είναι συστηματική ε, και στέρεα. Σε ό,τι αφορά τώρα την έλλειψη εναρμόνισης ε, μεταξύ του ουσιαστικού και του διαδικαστικού δικαίου ε, πρέπει να πω ότι εγώ θεωρώ ότι χάρη σε θεσμούς όπως η Eurojust και χάρη στο διάλογο μεταξύ ε, των δικαστικών μπορούμε να αποδεχθούμε τις, διαφορετικέ τις διαφορετικές νομοθεσίες. Η υπερβολική εναρμόνιση ορισμένες φορές κάνει κακό. Θα πρέπει λοιπόν ως κράτη-μέλη βεβαίως ε, να, ο καθένας να διαφυλάξει, να διαφυλάξει τη δική του ε, παράδοση ας πούμε την νομική αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Νομίζω πως είμαστε στο σωστό δρόμο. Χάρη στην Eurojust μπορούμε να έχουμε και διαφορές διότι μέσω του διαλόγου μπορούμε να ε, ξεπεράσουμε τις διαφορές αυτές. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Μπίλτσικ. Ε, η μετάβαση με τον νέο κανονισμό ε, είναι πρόσφατη αρχές Δεκεμβρίου. Ε, ξεκινήσαμε, είναι δύσκολο ακόμα να πούμε πώς θα μας επηρεάσει. Πάντως είναι θετικό ότι τα κράτη-μέλη τα οποία είχαν διαφορετικές προτεραιότητες ε, πλέον είναι στη Eurojust και αυτά ε, έχουμε και την Κομισιόν στο Δυτικό Συμβούλιο ε, νομίζουμε πως είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό τι άλλο Τέθηκαν δύο-τρία ερωτήματα σχετικά με το πολιτισμό νομικό πλαίσιο, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι ε, και γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο προπολογισμό μα. Ακούστε, πρώτα απ' όλα έχουμε όλο και πιο πολλέ υποθέσει που φτάνουν στα χέρια τη Eurojust. Όλο και πιο πολλά αιτήματα οικονομική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι διασυνοριακέ υποθέσει ε, είναι ακριβέ χρειάζονται μεταφράσεις, ε, χρειάζονται, χρειάζεται διερμηνία, χρειάζονται ταξίδια. Ε, οπότε οι εθνικοί προπολογισμοί δεν αρκούν για αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. Επίσης είναι όλο και πιο περίπλοκα τα πράγματα, ε, όλο και πιο πολλές διεθνείς υποθέσεις. Το νομικό πλαίσιο είναι όλο και πιο περίπλοκο, χρήζει διάλογο, διαλόγου, συνεδριάσει, ε, συντονισμού, έντονη συνεργασία. Ε, αυτά είναι που μας βοηθούν και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το καλό είναι ότι ο Επίτροπος μας υποστηρίζει και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χάμντραν, ε, ευχαριστούμε και όσους πήραν το λόγο. Εκτιμούμε την ευκαιρία που μας δώσατε ε, ευκαιρία που είχατε μάλλον να μας ενημερώσετε για τις προοπτικές ε, της Eurojust ε, και τις δυνατότητες μιας πιο, πιο αποτελεσματικής υποστήριξης. Ε, υπάρχει βέβαια το άρθρο της συνθήκης που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία και την πραγματογνωμοσύνη της Eurojust και ελπίζουμε ότι θα σας ξαναδούμε σύντομα Καθώς αποχαιρετούμε τον κύριο Χάμραντ, καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Ρέντερς Καλώς Yes, Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο 10 στην ημερησία διάταξη, λεγόμενο διαρθρωμένο διάλογο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Δικαιοσύνη, τον κύριο Ντιδιέ Ρέντεξ. Επ' θα μα ενημερώσει για τι δραστηριότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικό του χαρτοφυλάκιο που είναι το κράτο δικαίου. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, δικαστική συνεργασία, κυρίως σε ποινικά ζητήματα. και τα υπόλοιπα θέματα του χαρτοφυλακίου του. Θα γίνει και συζήτηση. Πρώτα ε, θα μιλήσουν οι συντονίστες και μετά θα υπάρχει χρόνος και για τα υπόλοιπα μέλη που θέλουν να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις αγωνίες τους για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Σηκώνονται κάρτες, σημειώνουμε τα ονόματα. Θυμίζω όμως ότι έχουμε προγραμματίσει τη συζήτηση αυτή μέχρι τις 12 παρατέταρτο, όπου έρχεται ε, η Κροατική Προεδρία για να μας παρουσιάσει τα δικά της θέματα και τις προγραμματικές της ε, δηλώσεις για το εξάμεινο. Καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καρά μου που ξαναέρχομαι ενώπιον της Επιτροπής σας, Επιτροπή Λίμπε, για να συζητήσουμε πολλά για την ιδιαίτερη κατάσταση σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, για το κράτος δικαίου. Ένα σας δώσω μια ευρύτερη εικόνα ε, του χαρτοφυλακίου μου σε σχέση με τη δική σας επιτροπή. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια ολόκληρη πλειάδα θεμάτων. Θέλω να συνεργαστώ πάρα πολύ στενά με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Το είπα ήδη αρχές Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Και ε, αυτές οι ανταλλαγές ε, απόψεων είναι καταπληκτική ευκαιρία να το κάνουμε. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι το κράτος δικαίου. Τα έχουμε συζητήσει αυτά επανειλημμένα. Είναι προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και για την αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, είναι αμοιβαίο υποφελώ και για την εσωτερική αγορά και για ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσει. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα συνολικό μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Η κυρία Φόντερ Λάιν μου εμπιστεύτηκε να ηγηθώ σε αυτή την προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συντονίζω το, την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου που θα καλύπτει τα διάφορα στοιχεία του κράτους δικαίου και ε, κυρίως συστημικά προβλήματα με ε, την έγκριση νομοθεσίας, ε, ελλειπή έλεγχος από ανεξάρτητα δικαστήρια, μη σεβασμός τη διάκριση των εξουσιών, η δυνατότητα των κρατών μελών και η ικανότητά τους να καταπολεμούν τη διαφθορά και όταν υπάρχει ε, διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ζητήματα πολυφωνίας του τύπου. Το 2016 στην έκθεσή σας εσείς ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα και τώρα θα θέλετε από ό,τι ξέρω να κάνετε και μια νέα έκθεση πρωτοβουλίας για να ενημερωθεί αυτό. Φέτος αρχίσουμε να εκδίδουμε την ετήσια έκθεση και ελπίζω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν συνέχεια. Πραγματικά θέλουμε να αρχίσουμε ένα άτυπο διοργανικό διάλογο έτσι ώστε να οικοδομηθεί αυτή η διαδικασία από κοινού, χωρίς αποκλεισμού και με επικοδομητικό πνεύμα. Ε, προσβλέπω στην υποστήριξή σας αυτή την προσπάθεια. Επίσης βασικό είναι ο διάλογος μας να επεκταθεί πέραν των Βρυξελών και να αρχίσει με τα εθνικά κοινοβούλια. Ελπίζω και πάλι σε συνεργασία μαζί σας να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη ε, διακοινοβουλευτική συνεργασία σε θέματα κράτους δικαίου. Αξιότιμα μέλη, θα πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι οι συζητήσεις για το νέο μηχανισμό δεν θα πρέπει να μας αποσπούν την προσοχή από κάποια ζητήματα και προβλήματα με το κράτος δικαίου σε κάποια κράτη-μέλη. Πρόσφατα συζητήσαμε και εδώ στην Επιτροπή σας και στην Ολομέλεια την κατάσταση στην Πολωνία, Ουγγαρία, Μάλτα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα έχω ήδη πει. Έρχομαι τώρα σε ένα σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται ε, διερεύνηση από το, την ποινική μας δικαιοσύνη και ε, προσαγωγή στην δικαιοσύνη των ε, ενόχων. Ε, μιλώ για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, ε, τον κανονισμό και τη σχετική οδηγία. Έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει το Κοινοβούλιο πώς έχει το χρονοδιάγραμμα και τι προτίθεστε να κάνετε ω επόμενα βήματα. Κατανοώ ε, τη θέση των διαφόρων πολιτικών ομάδων και φαίνεται αυτό με τι τροπολογίε που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Οι υπηρεσίε μου είναι στη διάθεσή σα για να αναλύσουν μαζί σα τι πρακτικέ ε, επιπτώσεις των διαφόρων εναλλακτικών ε, που υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι όμω στη δικαιοσύνη χρειάζονται επιγόντω ε, αυτό το εργαλείο και είμαι βέβαιος ε, πολλοί αγωνιούν να συνεισφέρουν και στη δική σας συζήτηση. Αντιμετωπίζουν ακόμα πολλές δυσκολίες όταν προσπαθούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές οι δυσκολίες δεν μπορούν να λυθούν ικανοποιητικά με τα σημερινά μέσα, εργαλεία και διαδικασίες που δεν είναι προσαρμοσμένα στο ψηφιακό κόσμο. Τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει με ειδικό τρόπο να αντιμετωπιστούν όπως ήδη γνωρίζετε δεχομένω, 27 ε, υψηλόβαθμοι ε, εισαγγελίε από τα κράτη-μέλη ε, προέβησαν σε δημοσίευση ανοιχτής επιστολής καταδεικνύοντας τις δυσκολίες της νομοθεσίας αυτής. Είμαι σίγουρος ότι ο στόχος είναι κοινό. Ας συνεργαστούμε για να βρούμε μια καλή και ισοπορεμένη λύση. Τα θύματα του εγκλήματος θέλουν να γνωρίζουν και επιθυμούν να γνωρίζουν ε, και το χρειάζονται ότι το ίντερνετ δεν είναι ένας χώρος ατιμορρησίας. Δεν μπορούν όλα τα θύματα ε, να ε, υπολογίζουν στα δικαιώματά τους. Γι' αυτό θέλω να έχουμε μια στρατηγική μέχρι το 2024 στην Ένωση για τα δικαιώματα των θυμάτων. Να υπάρχει μια σαφήνεια και μακροπρόθεσμα και να ενισχυθεί η σημερινή κατάσταση των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένε δράσει για την ενίσχυση τη συνεργασία και του συντονισμού για καλύτερη προστασία των πιο ευάλωτων θυμάτων, για διευκόλυνση τη πρόσβαση των θυμάτων σε αποζημίωση. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να έχει και μια εξωτερική διάσταση και να εξασφαλίζει περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες μας που πέφτουν θύματα αξιόπινων πράξεων σε τρίτες χώρες και να προωθεί τις αξίες γενικά στην ε, Ιφίλιο. Άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μένα. Υποστηρίζω απολύτως την κυρία Κοβέζη, την Γενική Εισαγγελέα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αρχίσει να λειτουργεί μέχρι τα τέλη του έτους. Επόμενο βήμα είναι ο διορισμός ε, του υπόλοιπου ε, των υπόλοιπων μελών από το Συμβούλιο για να μπορέσει να λειτουργήσει η εισαγγελία. Θα έχει στόχο να ε, εργάζεται με πολλές εθνικές νομοθεσίες και είναι σημαντικό να έχουμε προσέγγιση του ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα στο δικονομικό σκέλος. Ε, για να γίνεται σωστή η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξέδωσε εκθέσεις εφαρμογής για τις οδηγίες για τα δικονομικά ε, δικαιώματα η πράξη δείχνει ότι παραμένουν δυσκολίες σε βασικά σημεία των οδηγιών στην εφαρμογή τους. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, αποκοινούμε τα κράτη-μέλη, τους ενδιαφερομένους, ενεχομένους, τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις οδηγίες να είναι ουσιαστικά στην καθημερινή πρακτική. Είτε πρόκειται ε, ε, σε αστυνομικά τμήματα, είτε σε ε, δικαστήρια. Επίσης θα έχουμε και μια συνολική έκθεση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψη. Αυτό αναμένεται να εκδοθεί στα μέσα του έτους, φέτος. Και προσβλέπω και σε ε, έκθεση του Κοινοβουλίου που θα έρθει να και στο ρόλο του Κοινοβουλίου που θα είναι συμπληρωματικός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εντοπίσει τα κενά και τα ελλείμματα ε, στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Θα αναλύσω πολύ προσεκτικά τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και θα δώσουμε συνέχεια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ε, ως θεματοφύλακας των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, διστάζει στο να επιβάλλει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προσφεύγουμε και επί παραβάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσέφυγε κατά δύο κρατών μελών στο δικαστήριο και έχουμε επιβάλει και πρόστιμα ε, για τη μη μεταφορά ε, της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, με δύο άλλα κρατημέλη είναι καθοδόν η διαδικασία αυτή προσφυγής για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για να είναι ομοιόμορφη εφαρμογή. Το Μάιο θα εκδοθεί έκθεση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταβιβάσεις δεδομένων και τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Θα αξιοποιήσουμε και τις προτάσεις του Συμβουλίου, ε, του υπόπτη Προστασίας Δεδομένων και των άλλων ενδιαφερομένων. Βεβαίως, περιμένουμε να λάβουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, την πρότασή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης αυτό το καιρό ολοκληρώνει την αναθεώρηση που είχε αρχίσει η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς πρέπει να συντονιστεί καλύτερα το ποινικό δίκαιο με την προστασία των δεδομένων. Η νομοθεσία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε πολλούς από εσά και αποτελεί πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο. Με χαρά σας ενημερώνω ότι το Κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ε, ε, φέτος το Γενάρη ενέκρινε ένα νόμο που ενισχύει τις δυνατότητες επιβολής του νόμου του επόπτη δεδομένων. Όπως γνωρίζετε, μια ε, ανεξάρτητη εποπτική αρχή με δυνατότητες επιβολής του νόμου είναι προαπαιτούμενο για τη σωστή λειτουργία. Συνεργαζόμαστε με τους Κορεάτες αυτή τη στιγμή για να βρούμε λύσεις σε κάποιες διαφορές που απομένουν μεταξύ των συστημάτων μας, έτσι ώστε να ληφθεί ε, τους επόμενους μήνες απόφαση καταλληλότητας. Πριν τελειώσω, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα της τέχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα, πώς συνδέεται αυτή με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ένα σημαντικό τμήμα δευτερογενούς παράγωγου δικαίου εξασφαλίζουν την προστασία. Αλλά υπάρχει και το δεδομένο το θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, που επισκιάζεται από κάποιες σκοτεινές ε, πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης που ε, ξεφεύγει ε, του ελέγχου των κρατών μελών και ορισμένων δικαστηρίων επίσης. Θα πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές με βάση την εντολή τους. Όσο λιγότερο είναι ο έλεγχος ε, ανθρώπινο στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο έλεγχος και ευρύτερο. Και η προβλεψιμότητα θα πρέπει να είναι δεδομένη όταν ε, πρόκειται για εφαρμογέ που επηρεάζουν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι κοινέ οι ευρωπαϊκέ αξίε και μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό όταν τρέχουν οι εξελίξεις και χρήση των νέων τεχνολογιών. Χρειαζόμαστε μια σωστή καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται στις 19 Φεβρουαρίου να εκδώσει λευκή βίβλο με τα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος είναι ο στόχος? Να εξασφαλίσουμε ότι αυτή αναπτύσσεται με τις βασικές, παράλληλα με τις βασικές μας αρχές και αξίες και ε, βασίζεται στην ομοθεσία μας, στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο και προβλέψιμο για να μπορεί να λειτουργεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση. Ελπίζω αυτή η εισαγωγική μου παρουσίαση να σας έδωσε μια καλή εικόνα και επισκόπηση των προτεραιοτήτων που έχω ε, και για τη συνεργασία μας και, και βέβαια περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, τη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και που μας επικαιροποιήσατε για το θεματολόγιο σας σε σχέση με τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας. Καταρχήν ε, θα ακούσουμε τους συντονιστές και έχουμε και ένα μακρύ κατάλογο βουλευτών που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και να κάνουν σχόλια. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σεβαστείτε το χρόνο γιατί Στι 12 παρατέταρτο θα έρθει και η Κροατική Προεδρία. Δύο λεπτά παρακαλώ για τους συντονιστέ, έτσι ώστε μπορούμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπου ε, βουλευτέ. Η κυρία Μετσόλα για το έλεγχο καταρχήν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν ε, που αναλάβετε τα καθήκοντά σας και είστε τόσο αποτελεσματικός ε, τις πρώτες λίγες εβδομάδες και καθώς ε, η θητεία σας ε, θα χαρακτηριστεί από τη θέση λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ορόσημο μπορούμε να πούμε για τη δικαστική συνεργασία και την επιβολή του νόμου στην Ένωση. Είδαμε τις τελευταίες εκτιμήσεις από ε, την επικεφαλή εισαγγελία σε σχέση με τους πόρους που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ξεκινήσει και να καταστεί πλήρως λειτουργική. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκή προπολογισμό και ότι οι απαραίτητοι πόροι θα δοθούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ο πρόσθετος προϋπολογισμός που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, δεν θα δοθεί εις βάρος άλλων πρωτεοτήτων ε, στον τομέα της δικαιοσύνης. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσετε ότι η μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust μπορούν να συνεργαστούν ε, ως ομάδα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας ενώπιον αυτής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όταν παρουσιαστικό της υποψήφιος για αυτό το φάκελο, μας είπατε ότι θέλετε να συσταθεί ο μηχανισμός για το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου. Δώσατε κάποια στοιχεία στην αναρκτηριομιλία σας, αλλά μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η πρωτοενωμένη προθεσμία ε, ποιο είναι το προτεραιόμενο χρονοδιάγραμμα και ε, τι γίνεται με την ε, προθυμία, την έλλειψη προθυμίας που δείχνει το Συμβούλιο για να κινηθεί αυτό το θέμα στην προτεραιότητα. Κυρία Σίπελ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να επανέλθω και πάλι στο Brexit. Χθες είχαμε ένα σεμινάριο σε ό,τι αφορά την απόφαση επάρκειας και ξεπλάγει είναι που η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα αισιόδεξη με την αξιολόγηση πραγματεύσεις και τα πορίσματα ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του έτους, μου σε 11 μήνες μόνο. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα εξακολουθεί εξακολουθώντας να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομα αντέγραψε δεδομένα από το ΣΥΣ ε, και Μιλάμε για 75.000 τέτοια στοιχεία. Είπαν ότι ήταν τεχνικό πρόβλημα, αλλά ποτέ δεν ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση να ενημερώσω η γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των δεδομένων. Και θα έλεγα ότι ακόμη και η αρχή προστασία των δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν ικανοποιημένη για το πώ εφαρμόζεται ο Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων, κυρίω ό,τι αφορά τι εξαιρέσει σχετικά με την μετανάστευση, που μπορεί να οδηγήσουν ξεκάθαρα σε μεγάλα προβλήματα για του Ευρωπαίου πολίτε που παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι μέλος ε, του ε, δικτύου που λέγεται Five Eyes Spice. Πώς μπορείτε να είστε αισιόδοξου ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες μέχρι τα τέλη του έτους. Και πρέπει να διασφαλίσουμε επίση ε, ότι όλε οι διαπραγματεύσει ε, και τα αποτελέσματα αυτών με το Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν θα πρέπει να υποσκάψουν τα δικά μα πρότυπα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Λεχθέντων αυτών, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Λυπάμαι. Πολύ ωραία να προσφέρει να προσφέρεστε να επανέλθετε και να εξηγήσετε τι συνέπειε. Όμω, έχουμε συζητήσει επί μακρόλε συνέπειε και θα προτιμούσαμε η Κομισιόν να έχει κάνει από πριν αυτό το έργο. Προφανώ δεν κάνατε αυτή τη δουλειά, γιατί αναφέρατε την επιστολή κάποιων εισαγγελέων, αλλά έχουμε πολλού παίκτε, ακόμη και εισαγγελεί, ε, που δεν είναι ικανοποιημένοι 100% με την πρότασή σα, τουλάχιστον όχι όλοι. Ξέρουμε λοιπόν τουλάχιστον τη θέση σας, ξέρουμε ότι θα αγωνιστείτε για τη δική σας θέση. Επίσης, κατανοώ ότι ήδη μαζί με, τις πολιτικές, με κάποιες πολιτικές ομάδες ε, εδώ προσπαθείτε να ενισχύσετε τη δική σας θέση. Όμως ε, δεν θα πρέπει εσείς να κάνετε τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θα καθορίσουμε τη δική μας ε, θέση χωρίς τη δική σας συνεισφορά. Ε, και για το χρονοδιάγραμμα έχουμε το δικό μας χρονοδιάγραμμα και είμαι σίγουρη ότι θα παρακολουθήσετε τα πάντα, όμως δεν θα μας πείτε εσείς ε, πώς θα χειριστούμε τους διάφορους φακέλους. Ευχαριστούμε κυρία Ίντιβελ. από Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που ήδη ελέγχθησαν από τους συναδέλφους, την κυρία Μέτσολα και την κυρία Ζίπελ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την ανακοίνωση για την πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου, πρώτη της δικαίου, ως ε, εισηγήτρια ε, για το πακέτο αυτό. εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, πραγματικά όμως ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευθυγραμμίσει την έκθεση αυτή με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, να διευρύνουμε δηλαδή το πεδίο, να μην αφορά μόνο το θεσμικό κράτος δικαίου, αλλά όλα τα στοιχεία του άρθρου 2, δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, όλα αυτά ε, είναι αδιάρρηκτα μεταξύ τους. Ε, επίσης, συστάσεις αναχώρα, να μην βασιζόμαστε μόνο σε πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις εθνικές κυβερνήσεις για προφανεί λόγους. Ε, ε, επίσης, η έκθεση καλό είναι να οδηγήσει μια συζήτηση όχι μόνο εδώ, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια και στο Συμβούλιο, διότι όπω είπε η κυρία Μέτσολα, είναι σημαντικό να συμμετάσχει και το Συμβούλιο ε, και θέλει λίγο πίεση εκεί. Ένα άλλο γενικό σχόλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει και η ίδια να σέβεται το κράτο δικαίου και υπάρχει μια τάση στην προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι εξ αυτήν, υπάρχει μια τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοείται παντελώ αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Και κοινικά περιμένουν από του πολίτε ε, να προσφύγουν. Ε, Είπε υπόθεση τη πράγματι Σίλ και ο κύριο Ρήμ, όπου έπρεπε να έχει κάνει τη δουλειά τη η Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να επαγρυπνείτε όταν οι συνάδελφοί σα ε, υποβάλλουν προτάσει που δεν σέβονται ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, Τέλο, για την ε, προστασία δεδομένων, είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι θα ε, ανανεώσετε τα εργαλεία προστασία δεδομένων τρίτου πυλώνα, του πρώην τρίτου πυλώνα, και η εφαρμογή του GDPR ε, είναι ανεπαρκής. Αυτό νομίζω είναι όλο και πιο σαφές ε, και αυτό σχετίζεται βέβαια με το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι αρκετά άτολμη ε, η προσπάθεια που γίνεται. Πώς το βλέπετε αυτό και πώς βλέπετε και το GDPR σε σχέση με το Brexit. Ευχαριστώ. Ναι, σας θυμίζω, παρακαλώ δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σας ε, για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Είναι και πολλοί αυτοί που θέλουν να μιλήσουν, ε, να έχουν όλη την ευκαιρία να παρέμβουν, να απευθυνθούν στον κύριο Ρέιντερς, ε, αλλά να μπορείς και ο ίδιος να έχει το χρόνο να απαντήσει. Και τώρα περνάμε στην κυρία Στρίκ για τους πράσινους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και Reinders για την ε, παρουσίαση ε, και που είστε εδώ βέβαια. Χαίρομαι που μας λέτε ότι θα ε, εφαρμόσετε αυτή τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. αναμένουμε την πρώτη ετήσια έκθεση βέβαια και αναμένουμε να δούμε πόσο συγκεκριμένες θα είναι οι πληροφορίες, γραπώς θα λαμβάνουν υπόψη και πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές. Ε, είμαστε περίεργοι λοιπόν να δούμε πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκές επίπεδων εξαρτησίας σε ό,τι αφορά τις πηγές των πληροφοριών επί των οποίων θα βασίζετε την έκθεσή σας. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο από αυτού, θα ήταν χρήσιμο. Ποια θα είναι δηλαδή η μέθοδος που θα ακολουθήσετε. Θα γνωρίζετε ότι εμείς ε, θα θέλαμε ε, πιο φιλόδοξα βήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ενός πιο ε, συνολικού μηχανισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια της διαδικασίας και που να περιλαμβάνει διαφορετικά κίνητρα από την πρόληψη έως και βεβαίως το άρθρο 7 που είναι το ίστατο μέτρο. Θα θέλαμε να ξέρουμε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο μηχανισμό. Θα υπάρξουν περισσότερα κίνητρα. Πώς θα αξιολογήσετε τις αιτήσει εκθέσεις εάν χρειαστούν περαιτέρω ε, μέτρα μετά από αυτή την αιτήσια έκθεση. θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση των κρατών μελών ή πρέπει να πάμε παραπέρα. Επίσης, για το άρθρο 7, το επίπεδο, το, η έλλειψη μάλλον πολιτικής βούλησης δυσκολεύει τα πράγματα σε επίπεδο Συμβουλίου. Ε, η Κομισιόν ε, νιώθει ότι υποστηρίζεται ότι θα είναι τα πρώτα ε, χρησιμοποιώντας άλλα μέσα ε, όπως ε, κάποιες προσφυγές μεταξύ χωρών για χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται συστηματικά με το κράτος δικαίου και τελευταίο ερώτημα για την αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη στην ποινική συνεργασία υπάρχει εδώ ο κίνδυνος επιδίνωσης του κράτους δικαίου και σχετικών προτύπων και αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη συναρμόνιση ό,τι αφορά τις ε, ε, δικλείδες ασφαλείας, τα εχέγγυα ε, τα διαδικαστικά σε υψηλότερο επίπεδο. To ID, Honorable Tardino, is she here? No. Είναι εδώ η κυρία Τερντίνο από το ID, όχι. Τότε να περάσουμε στον επόμενο συντονιστή, ο κύριος Γιάκη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Θα ήθελα Καταρχήν ε, να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε στις ε, ηλεκτρονικές αποδείξεις. Είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά μπορούμε ε, να ξεκινήσουμε από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Επίσης, ε, υπενθυμίσατε πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τμήμα των καθηκόντων Σα επομένω, θέλω να σα ρωτήσω πόσο ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και συγκεκριμένα την περιθμό 12 που λέει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα να συνεταιρίζεστε και ελευθερία της έκφρασης πώς ε, αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα γίνεται σεβαστό στη Γαλλία. Πριν ε, κάποιες εβδομάδες ε, διαδήλωσαν κάποιοι εργαζόμενοι στη δικαιοσύνη και ήταν θύματα βίας στο δρόμο και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο αν σκοπεύει να κάνει κάτι σχετικά με αυτή την παραβίαση ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συνθήκες ισχύουν ε, για όλα τα κρατημέλη, κάποια τελικά είναι πιο ίση από άλλους. Και από τη Σκοπιά της Πολωνίας έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 κατά της Πολωνίας ε, θα υπάρχει μια ψηφοφορία, υπάρχει επαρκής πλειοψηφία ε, για το θέμα αυτό σύμφωνα με τις συνθήκες. Γιατί μέχρι τώρα φαίνεται ότι η υπάρχουν κάποιες κατηγορίες σχετικά με πολιτικές παρεμβάσεις στο δικαστικό τομέα για το πώς εκλέγονται οι δικαστές στην Πολωνία, σε άλλες χώρες όπου υπάρχει πολιτική εκλογή των δικαστών. Τι γίνεται, θα αναλύσει η Κομισιόν αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε όλες χώρες όπου δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Η κυρία Έρνστ. Από την Ενωτική Αριστερά, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω ε, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Σημαντικά όλα αυτά και για μας, δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι το θέμα του κράτους δικαίου ε, κυριαρχεί και είμαστε πολύ περίεργοι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Περιμένουμε, έλεγα επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον την ετήσια έκθεση. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό, το έχουμε ξανασυζητήσει για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Και συστάσεις αναχώρα να κάνετε. Γιατί όχι. Αλλά εντάξει, οι συστάσεις είναι συστάσεις. Πώς εφαρμόζονται. Καλό είναι να απευθύνει συστάσεις, αλλά αν δεν προχωρήσουμε πρέπει να, σταματήσουμε να συζητάμε για άλλα νομοθετικά εγχειρήματα και ε, σχέδια. Αφού έτσι και τα κράτη-μέλη δεν τα εφαρμόζουν ή τα εξουδετερώνουν τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Συμφωνώ με τους εισηγητές. Ε, ήταν σαφής η θέση τους. Και εμείς ως πολιτική ομάδα πιστεύουμε ότι είναι επίμαχο το κατά πόσο είναι ε, σκόπιμη και λογική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα μας το αμφισβητεί αυτό. Τελευταίο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων συζητούμε την εφαρμογή σε βάθος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα κράτη-μέλη στην εφαρμογή, γιατί εμεί θέλουμε να υπάρχει ομοιόμορφη, ενιαία. Και να μην έχουμε ελλείμματα ή διαφορές στην προστασία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θέλω απλώς έκθεση εδώ, αλλά και συμβουλές να δίνετε και συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τα σημειώσατε όλα αυτά. Εδώ και ώρα βλέπω να σημειώνεται. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Να ακούσουμε και τους υπολείπους για να απαντήσετε εσείς στο τέλος. Έτσι πιο συνολικά. Για οικονομία χρόνου. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παραβιάσουμε το χρονοδιάγραμμά μας και δεν θα πάρουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι. Παρακαλώ να τηρείτε και εσείς το χρόνο σας έχετε στο μυαλό σας. Ένα λεπτό, ένα άμεση το πολύ, για να μπορέσει να απαντήσει με την ησυχία του ο Επίτροπος, γιατί έχουμε 20 και πλέον συναδέλφους. Ο κύριος Χετβέγγι. Ευχαριστώ. Μου δώσετε το λόγο νωρίτερα από την νόμιση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το, σημαντικό σας, ε, το σημαντικό σας έργο. Καλή τύχη. Θέλω να μιλήσω για το θέμα του κρατούς δικαίου. Πρόκειται για έναν ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατιών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά την ίδρυσή της. Και κάποιοι βασικοί πυλώνες ε, είναι το να υπάρχει αντικειμενικότητα και οι κανόνες για όλους και όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επίσης, να βλέπουμε ποια είναι τα γεγονότα. Τώρα, η κριτική μας για το τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι υπήρξε έλλειψη αντικειμενικότητας ε, και για πολιτικού και ιδεολογικού λόγους υπήρχε κατάχρηση. Και αυτό δεν αντίκειται μόνο στο κράτος δικαίου, αλλά και στη σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και υποβιβάζει την ίδια την έννοια. Βλέπω την δραστηριότητα του Επιτρόπου Τίμερμανς ε, περισσότερο σαν ένα παρτιζάνο παρά ως αντικειμενικό παίκτη στον τομέα. Πώς θα διασφαλίσετε εσείς ότι η αντικειμενικότητα θα γίνει βασικό μέρος της συζήτησης για το κράτος δικαίου και σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες τις οποίες βασίζονται η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι είναι ισορροπημένες οι πληροφορίες και αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα και όχι πολιτικές εκστρατείες. Κύριε Μπάρλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ εγώ θέλω να αφαιρθώ στο κράτος δικαίου βεβαίως. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά ένα κράτος μέλος στην Πολωνία. Έχουμε δει αποκαλούμενες 30 μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρωτοφανές. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ε, ουσιαστικά προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά τμήματα γιατί έχουμε δει πολλούς ε, προβληματικούς ε, κανόνες. Ποιες ε, προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται πριν να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πόσο μπορεί να περιμένει η Κομισιόν σε τέτοιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι δυνατόν να προσφύγει σε πρώιμο στάδιο, μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Μπάρλι. Κυρία Κύριο συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτρο που είστε εδώ και απαντά τι ερωτήσεις μας. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω και τη δουλειά σας ε, για το κρατός δικαίου, τις σχετικές εκθέσεις και ότι θα παρουσιάσετε ήδη φέτο ε, τι πρώτες. Πολύ καλά ήταν αυτά. Και φυσικά έχετε την υποστήριξη της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου για το θέμα του κράτους δικαίου και το σχετικό μηχανισμό γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, αλλά να δείξουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι προστατεύουμε τα δικαιώματά τους και προστατεύουμε τη δημοκρατία και ότι αυτό αποτελεί βασικό μέρος του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εμείς στο Κοινοβούλιο θα απευθύνουμε έκκληση ο μηχανισμός αυτός ε, να εγγραφεί σε μια διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων Φυσικά καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας για τον άτυπο διάλογο μεταξύ των οργάνων, αλλά θεωρούμε ότι ο ίδιος ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι προβλέψιμος, νόμιμος και νομικά δεσμευτικός μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας. Έχω και ένα ακόμη σχόλιο και ερώτηση. Το σχόλιο, είπατε κι εσείς, ότι αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της διαδικασίας του άρθρου 7, αλλά θα είναι κάτι συμπληρωματικό. Και Κάτι τελευταίο για τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Πώς βλέπετε το σύνδεσμο μεταξύ αυτού του κανονισμού και την ερεσιμότητα για το κράτος δικαίου και του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων επί του οποίου εργάζεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ζαζραήλ. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομος και ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να φύγω λόγω της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς βλέπετε την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα αξιολογεί το κράτος δικαίου. Διότι ε, κάτι που δεν λειτουργεί και τόσο καλά ε, στα πλαίσια του άρθρου 7 είναι ότι επικεντρωνόμαστε σε κάποιες επιμέρους χώρες με έναν τέτοιο τρόπο που δεν ε, διαφυλάσσει ουσιαστικά την αξιοπρέπεια της χώρας αυτής και του λαού της χώρας αυτής. Αν υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, δίκαιος, αμερόληπτος για τα 27 κράτη-μέλη, ε, νομίζω ότι έτσι θα αποφύγουμε αυτήν την, ε, αυτόν το, αυτήν τόσο, την όχι τόσο δίκαιη αξιολόγηση. Ε, Λοιπόν, ποια είναι τα βήματα που σκοπεύει να ε, κάνει η Κομισιόν έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο μόνιμος μηχανισμός. Ευχαριστώ. Κανίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να σας θέσω μια ερώτηση πάντοτε σε σχέση με την ενίσχυση του κράτους δικαίου από διαφορετικό προφίλ όμως γιατί θεωρώ ότι το κράτος δικαίου σήμερα απειλείται από κάποιες μορφές εγκληματικότητας, π.χ. η τρομοκρατία, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα. Και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα. Έτσι όπως έγινε και στην προηγούμενη θητεία σε σχέση με την τρομοκρατία, μήπως θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος με μια ενωπημένη στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι σε μια νομοθεσία που παραδείγματο χάρη να υπερβαίνει τις ε, νομοθετικές διαφοροποίησεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Ακούσαμε πριν τον πρόεδρο της, ε, του διευθυντή της Eurojust που μας είπε ότι χάρη στην ε, συνεργασία που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και χάρη στο έργο της Eurojust μπορούν να καλυφθούν κάποια από αυτά κενά. Όμως ε, έχουμε διαφοροποιημένες νομοθεσίες που δημιουργούν νομοθετικά κενά που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες. Σας ρωτώ λοιπόν μήπως θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ομοιόμορφη που να ξεκινά από έναν ενιαίο ορισμό του οργανωμένου κλίματος ε, και να ε, υπερβαίνει τα προβλήματα που έχουμε στον κανονισμό 841. Επομένω, μήπω να δούμε πώ θα εναρμονίσουμε την νομοθεσία στον τομέα αυτό. Επίση, σα ευχαριστώ ε, που απαντήσατε ήδη ε, σε μία ερώτηση που θα θέτω εγώ για τη θέση σε λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ, κυρία Παχασαρτουνδουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με το έργο τη κυρία Κινίτσι. Το οργανωμένο έγκλημα έχει μεταλλαχθεί και πρέπει να το ενεργοποιήσουμε με πλουσματικό τρόπο διότι τελικά αποτελεί απειλή για την ακαιρεότητα της δημοκρατίας σε κάποιες από τις χώρες μας. Και δύο ακόμα ερωτήματα. Ένα για το πακέτο που, που έχει να κάνει με τα θύματα. Ε, θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτό που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή η οποία είναι εξαιρετικά ελληματική της οδηγίας του 2012 για τα θύματα ε, οποιαδήποτε μορφή εγκλήματος πρέπει να λαμβάνετε υπόψη εδώ. Φαντάζομαι ότι επίσης ότι θα λάβετε υπόψη σας και αυτά που λέει το άρθρο 2017 στο, για τις τρομοκρατικά εγκλήματα και τα θύματα. Κατά πώς θα λάβετε υπόψη λοιπόν τις συστάσεις της ειδική Επιτροπής για την Τρομοκρατία του 2018 που γίνεται ε, ε, ρητή αναφορά στο να αποφύγει να η διπλή θυματοποίηση ε, δηλαδή να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί αλλά κυρίως να μην γίνουν θύματα και δεύτερη φορά και το, το, επόμενο ερώτημα μου έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να στραφεί κατά των, των ανθρώπων, κατά των θεμελιών δικαιωμάτων τους. Αναφερθήκατε στο θέμα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα να ξέρω πώς περιλαμβάνεται εδώ τη δυνατότητα νομοθεσίας ε, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση ε, προσώπου. Ο κύριε Μπίλτσικ, ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω ε, και τον Επίτροπο Ρέιντερς για την ανταλλαγή απόψεων. Έχετε βάλει στην πρώτη γραμμή, βλέπω, των προτεραιοτήτων σας το ζητήματα κράτους δικαίου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχω κάποια ερωτήματα. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρωτοβουλία να δημοσιεύονται οι αιτήσεις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, να θευτεί από επιτυχία και να οδηγήσει τελικά σε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο για το κράτος δικαίου με όλα τα θεσμικά όργανα. Αυτό θα ήταν κάτι που θα μας βοηθούσε, πιστεύω. Γι' αυτό θέλω να αφαιρθώ και στο πεδίο και τη φιλοδοξία ουσιαστικά αυτής της πρώτης έκθεσης ε, που θα δημοσιευθεί είναι ένα πρώτο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημά μου είναι θα δώσετε έμφαση στην πρόληψη, ε, θα εξετάσετε όμως και κάποιε κάποιες με βάση βεβαίω τα ευρήματα και τις αξιολογήσει που θα προκύψουν. Και κάτι άλλο, επειδή είναι εξαιρετικά πολιτικό το ζήτημα, οπότε θα αποτελέσει μέρος και του πολιτικού διαλόγου. Ε, ποια θα είναι η επικοινωνιακή σας στρατηγική ενώπιση των εκθέσεων αυτών έτσι ώστε να προλάβουμε τις κριτικές, ε, τις αντιδράσεις ε, των ε, σκεπτικιστών είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο το τι δημοσιεύουμε αλλά και το πώς το πλαισιώνουμε πώς επικοινωνούμε γύρω από αυτό έχετε κάποια στρατηγική γι' αυτό ε, ευχαριστώ κυρία Γιόντσεβα έχει το λόγο ευχαριστώ πρόεδρε ευχαριστώ κύριε Πίτρο για τις πληροφορίες θέλω να πείτε την προσοχή σας σε ένα στοιχείο του κράτου δικαίου, του σχετικού μηχανισμού, την αντιμετώπιση τη διαφθοράς. Εδώ και χρόνια οι προκλήσεις ε, που μας ε, θέτει η διαφθορά σε διάφορα κράτη-μέλη υποτιμώνται. Είναι λίγα και τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει μια σφαιρική στρατηγική αντιμετώπιση τη διαφθοράς. Αντιλαμβάνομαι ότι η αντιμετώπιση τη διαφθορά είναι ένα δύσκολο ζήτημα Πολλοί, θέλουν να αποφύγουν ένα τέτοιο ευαίσθητο τοξικό ζήτημα. Είμαι από τη Βουλγαρία, όπου η διαφθορά πραγματικά κάνει μεγάλη ζημιά σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτό δημιουργεί και ευρωσκεπτικισμό. Είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη και ξέρετε ότι η αλυσίδα, η αλυσίδα έχει τη δύναμη του πιο δύναμου κρίκου της. Ε, έχω δύο ερωτήματα για σας. Ε, θα υπάρξει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ε, διαφθοράς όχι μόνο στα πλαίσια του κράτους δικαίου, αλλά ως μια αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική. Και τι είδου μέτρα, τι είδου προτάσει μπορούν να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη διαφθορά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή, εφόσον ελέγχθη ότι δυστυχώ η ομάδα τη εισαγγελέα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων. Μάλιστα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ και καλή τύχη για το έργο σας στην επόμενη περίοδο. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, η πρώτη σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι έθεσαν σχετικές ερωτήσεις. Είναι όμως προτεραιότητα αυτή τη επιτροπή και χαίρομαι που ακούω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η προηγούμενη ε, Κομισιόν ε, σημαντικά υποτίμησε τις ανάγκες ε, στελέχωσης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και το θέμα της χρηματοδότησης. Μόνο 32,5 εισαγγελίες είχαν προβλεφθεί για περίπου 900 υποθέσεις και μόνο η Ρουμανία έχει περίπου 900 συνεχιζόμενες υποθέσεις απάτης αιτησίως, που αφορούν ευρωπαϊκό κονδύλια και έχουμε πολλούς εισαγγελίες που εργάζονται σε αυτές τις υποθέσεις. Έχετε ε, κάποιες πρόσθετες, πρόσφατες εκτιμήσεις ε, για τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία των αναγκών της ΕΠΑ και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και η δεύτερη ερώτηση είναι πώ θα δώσουμε πιο συντονισμένη απάντηση απέναντι ε, στην καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων, ε, του οργανωμένου εγκλήματος ε, και τη νομικής παράνομων εισόδων. Δεν αρκούν τα όσα κάνουμε. πώ θα αντιμετωπίσετε αυτά και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στομπέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και καθώς ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έχω μια ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες των κρατών μελών να λάβουν αποφάσεις ε, για την απέλαση καταδικασθέντων εγκληματιών. Γιατί βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη ξενόμενη δραστηριότητα, έχουμε διασυνοριακές συμμορίες που εκμεταλλεύονται την ελευθερία της κυκλοφορίας και φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Και σε ό,τι αφορά αυτές τις εγκληματικές συγχωρίες, ε, όταν διαπράττουν πολύ σοβαρά δικήματα, φυσικά έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε αποφάσεις για πέλαση, όμως ε, πολλές από αυτές τις συμμορίες επικεντρώνονται, περίπτωση χάρη, σε διαρρήξεις και μπορεί να καταδικαστούν. Και κατόπιν ε, βλέπουμε ότι το σημερινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά πολύ δύσκολο το να ληφθούν αποφάσει απέλαση αν ε, είναι η υπήκοη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τον υπήκοη τρίτη χώρα η Κομισιόν σκοπεύει να λάβει πρωτοβουλίε ε, για να το διευκολύνει αυτό. Γιατί έχω ε, αυτό το πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στη Σουηδία, στη χώρα μου, έχουμε περίπου 70% όλων των διαρρήξεων που διαπράττονται από τέτοιε εγκληματικέ συμμορίε. και φυσικά προσπαθούμε να απαντήσουμε μέσα στην νομοθεσία μας, τους καταδικάζουμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να του στείλουμε πίσω στη χώρα του. Γιατί είναι υπήκοοι κράτου μάλιστα Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πουρίκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, έχουν περάσει 25 μήνε από το που ενεργοποιήθηκε η διαδικασία επί το άρθρο 7 κατά τη Πολωνία. Δυστυχώ δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, είναι ακόμη χειρότερη. Ε, καθώς η κυβέρνηση έχει λάβει πρωτοβουλίες ε, κατά ε, του δικαστικού σώματος. Έγινε και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα και την Πέμπτη διευθυντή ένα σημαντικό ψήφισμα σε σχέση τώρα με την ε, προσφυγή ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα γίνει στη συνέχεια και ποιο, τι γίνεται με τον ε, μηχανισμό, θα ενισχυθεί με περαιτέρω κονδύλια, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα ενισχύσουμε τις τοπικές αρχές και άλλους άμεσους δικαιούχους κατά των αποτελεσμάτων αυτού του μηχανισμού και αν θα είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι ευρωπαϊκέ συνθήκε ε, και αυτό το μηχανισμό προκειμένου να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σαρσαλέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την άδεια των συναδέλφων, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίασή σας και για τα όσα επί της ουσίας μας προτείνεται. Είναι πάρα πολύ απαραίτητη η συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο για να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας. Να λειτουργούν σωστά τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα και να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του εγκλήματος ε, για να είναι πιο ασφαλής η Ευρώπη. Υποστηρίζω θερμά την ανάπτυξη αυτού του νέου μηχανισμού που μας εξαγγείλατε, το μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Επειδή οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους, ε, Ελπίζω να ξανάρθετε στο Κοινοβούλιο και να μας εξηγήσετε σε λεπτομέρειες όλη τη διαδικασία και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Είναι σημαντικό κατά την απόψη μου. για να απαντήσουμε σε ένα αίτημα της κοινή γνώμης. Αναφερθήκατε στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Το έχουμε μελετήσει αυτό το θέμα, ιδιαίτερα την έκθεση, ε, με την έκθεση εφαρμογή. Και ελπίζω να μπορέσετε εσείς να βασιστείτε στα όσα πετύχαμε εμείς που είναι αρκετά για να οικοδομήσετε πάνω σε αυτά και να τελειοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο μηχανισμός. να φτάσει στο στόχο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κελέγα, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Ρεντέρς, όπως είπε και η συνάδελφος Ραμόνα ε, Στρογκάριου, καλή τύχη. Έχετε όλη την υποστήριξή μας. Τώρα έχετε ανασκουμποθεί και έχετε μπει ε, στην ουσία των υποθέσεων και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, για να προωθήσετε τα θέματα. Οι συνάδελφοί μου τα ανέφεραν προηγουμένως. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη δικαστική συνεργασία. Προηγουμένως είχαμε εδώ το Eurojust που εντάξει καλά δουλεύει, αλλά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Δεύτερον, στην επιστολή, ανάθεση αποστολή σας, η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν σας ζήτησε να φροντίσετε η δικαστική πολιτική εγκάρσια να καταπολεμά την ε, τρομοκρατία, τον εξε, εξτρεμισμό και να προαγάγει την ασφάλεια. Αυτό το θέμα δεν το θίξαμε πάρα πολύ. Ε, κατά τη διάρκεια της ε, προεκλογικής εκστρατείας, εμείς είχαμε ζητήσει μέχρι και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού FBI. Οι πολίτες περιμένουν περισσότερη αποτελεσματικότητα. Οι κακοποιοί και οι εγκληματίες εδώ και καιρό έχουν καταλάβει πώς ε, μπορούν να ε, χειραγωγούν και να φέρουν απέναντι ε, το ένα δικαστικό ή αστυνομικό σύστημα με το άλλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Πελτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Εγώ ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση των ευρωπαϊκών φυλακών που είναι πολύ ε, φρικτή και πώς διαβιούν οι κρατούμενοι. Στην Πορτογαλία 106 θέσεις για 100, 115 στην Ιταλία, 120 στη Ρουμανία, και αντίστοιχα είναι τα στοιχεία και στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ε, τακτά χρονικά διαστήματα καταδικάζει τα κράτη-μέλη για συνθήκες κράτησης που παραβιάζουν ε, το άρθρο 3 ε, του σχετικού τη Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το 2019 το Δεκέμβριο καταδικάστηκε η Πορτογαλία, δύο μέρε αργότερα η Γαλλία. Δέκα χώρε αρνούνται να εκτελέσουν ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Τι θα κάνετε για ενισχύσετε τα δικαιώματα των κρατουμένων και την πρόσβασή τους στα δικαιώματα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ε, στη δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την ενημέρωση και για την παρουσία σας. Έχω μια ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως αναφερθήκατε στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο γεγονός ότι το Φεβρουάριο θα έρθει η Λευκή Βίβλος. Πριν από λίγους μήνες επίσης ε, είπατε ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο ε, οριζόντιο και κάθετο. Αυτό παραμένει ή έχει καταργηθεί σε αυτό που θα προτείνετε το Φλεβάρι. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούν και Χόνσταϊν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Δηλώσατε προθυμία για συνεργασία. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας. Στους καιρούς που ζούμε, το δικό σας χαρτοφυλάκιο και εκείνο της κυρίας Γιώροβα είναι τα σημαντικότερα για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε σε διάφορα ζητήματα. Το, το διαδίκτυο δεν είναι χώρος ατιμορρησίας, είπατε. Επίσης, μιλήσατε για τα δικαιώματα των θυμάτων και την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζετε ότι υπάρχουν μαζικές εκστρατείες ρητορικής μίσους και κατασυκοφάντησης, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Και συχνά δεν στρέφονται μόνο απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους στην αντιπολίτευση, αλλά και κατά δικαστών. Είχαμε μια καμπάνια που ξεκίνησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πολλές φορές στρέφονται κατά υψηλά ισταμένων προσώπων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, άλλων και ε, συνοδεύονται από μαζική εκστρατεία παραπληροφόρησης. For Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, θυματοποιεί κόσμο, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζει κάμια στρατηγική κατά του φαινομένου αυτού, το οποίο διονγκώνεται συνεχώς. Το ρωτώ και στα πλαίσια της Λευκής Βίβλου που μας ανακοινώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now we have completed... Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε έναν αρκετά μεγάλο κατάλογο ομιλητών. Κύριε Επίτροπε, με σημειώσατε. Ναι, βέβαια, σας βλέπω. βλέπω ότι ζητάνε και άλλοι το λόγο. Ναι, να ακούσουμε ακόμα κάποιες ε, παρεμβάσεις. Παρακαλώ, κύριε Τοντοράτσε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγία για τα θύματα, στην οποία, την οποία ανακοινώσατε το 2024, αν κατάλαβα καλά, δεν είναι ακριβώ και πυροτέχνημα να μας λέτε ότι θα κάνετε κάτι το 2024 γιατί αργεί ε, τόσο πολύ. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνετε όλα στην αρχή βέβαια, αλλά τελευταία έτος τη θητείας, ε, τι να πω, μπορεί να με κατάλαβα καλά. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να προσθέσω κι εγώ στα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με του πόρου. Από ό,τι κατάλαβα, και πάλι ελπίζω να κατάλαβα καλά, για την ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ε, στη δημοσιονομική γραμμή. Ε, οπότε υπάρχει ένα στους ανταγωνισμού έτσι, με άλλες υπηρεσίες, με άλλους οργανισμούς. Ποιος είναι πιο σημαντικός, Europol, Eurojust, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο. Πρέπει να είναι με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λοιπόν. Ε, εκτός αν δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά. Ενδεχομένω από κοινού τον κύριο Χάν να το διορθώσετε αυτό. Τρίτον, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Θα είμαι σύντομο. Ξέρω ότι θα έχουμε την, ε, τη Λευκή Βίβλο. Πέρα όμως από τα λόγια ότι θέλουμε ανθρωποκεντρική προσέγγιση και προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, πώς θα βρεθεί το σημείο ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης ε, της πρόθεσης της καινοτομίας ε, έτσι ώστε να είμαστε όντως στην πρώτη γραμμή παγκοσμίω ε, στην τεχνητή νοημοσύνη ε, και αφετέρου να προστατεύσουμε τα ηθικά πρότυπα. Ποια διαφοροποίηση θα μας βοηθήσει να βρούμε αυτή τη λύση, αυτό, αυτή, το σημείο ισορροπίας. Θα γίνει κάποια αξιολόγηση κινδύνου. Ε, και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό που είπε ο πρόεδρος της Eurojust νωρίτερα ότι τα ηλεκτρονικά στοιχεία, ε, παιδιτικά στοιχεία δεν είναι απαραίτητα ένα σημαντικό εργαλείο ε, στο πλωστάσιο. Εγώ νομίζω ότι είπατε το αντίθετο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κλείνει ο καταλόγος τώρα, ε, δεν θα μπορέσει ο επίτροπο ε, να ε, μπορέσει πραγματικά να κάνει δομημένο διάλογο όπως ονομάζεται αυτή η διαδικασία. Κύριος, ο κύριο Κιόρνερ, μετά ο κύριο Μπράιερ και μετά η κυρία Πλησνιεύσκα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι σας ενδιαφέρει το θέμα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, εμείς ε, ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθούμε στενά το θέμα αυτό. Είναι ένα εργαλείο που είναι φιλοευρωπαϊκό θα έλεγα, αλλά χρειάζονται και κάποιε δικλείδε ασφαλεία σε των μελών δικαιωμάτων και ψάχνουμε μια συμβαστική λύση από αυτού. Ε, ένα ερώτημα όμω, διότι τα ηλεκτρονικά πολιτικά στοιχεία είναι το σημείο αφετηρία για τι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ. Ενδεχομένως να μπορείτε να μας πείτε κάτι για τις προγραμματεύσεις με τους Αμερικανούς ε, και ενδεχομένως επίσης ε, αν μπορείτε να μας αξιολογήσετε τη συμφωνία ε, των, των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο μιας και το Ηνωμένο είναι ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι η θέση σας επ' αυτού Ευχαριστώ ο κύριος Μπράιερ Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ένα θέμα ήθελα να θίξω γίνονται κάποιες συζητήσεις για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει ένα μορατόριο σε ό,τι αφορά την αναγνώριση προσώπου για λόγους παρακολούθησης. Είναι κάτι που συζητείται λόγω ε, το, το πόσο πραγματικά ε, εντυπωσιακό είναι η εντυπωσιακή αυτή τεχνολογία και το πόσο αδιάκριτα μπορεί να ε, έχει επιπτώσει του ανθρώπους του να μπορεί δηλαδή να σκανάρει πλήθη και να αναγνωρίζει πρόσωπα. Ε, ναι, η κυρία Βυσνιεύσκα τέλος. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν είναι μόνο το οργανωμένο έγκλημα, είναι και η διαφθορά και αυτό πρέπει να κυριαρχήσει ε, στη σκέψη μας και στη δράση μας. Παράδειγμα, η Πολωνία πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε κατά πολέμηση της διαφθοράς, έκλεισε ε, το έλλειμμα που υπήρχε στο ΦΠΑ και ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, πάνω από 260 δισεκατομμύρια σλότη. Άλλο θέμα είναι ε, η ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε, το ξέπλυμα κοινος και η απέλαση έκδοση των εγκληματιών. Είπατε ότι θέλετε να προστατεύσετε το κράτος δικαίου. Πώς προτίθεστε να το κάνετε αυτό συγκεκριμένα. Και επίσης ερωτώ κάτι για το άρθρο 7 της συνθήκης. Η ένομη τάξη και το πώς αυτή διαμορφώνονται είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Και θα σας παρακαλέσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, ε, υπερβαίνει τις συνθήκες. Είναι και θεματοφύλακα των συνθήκων. Ε, διαφωνώ με αυτό που είπατε και με τη διαδικασία για τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις στην Πολωνία υπάρχει τρομερή παραπληροφόρηση. Θα έχετε πολλή δουλειά και εδώ στην Επιτροπή μας και γενικότερα. Γιατί πολλά ακούσαμε και εδώ που είναι παραπληροφόρηση. Παρακαλώ να μην χειραγωγηθείτε πολιτικά, μην πείτε σε αυτό το παιχνίδι. Όλα τα θέματα τα οποία θίξατε σχολιάστηκαν πάρα πολύ από ε, τους βουλευτές, κυρίως συνδικαστική συνεργασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ε, κατά της μαφίας, διαφθοράς, ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολλά λοιπόν έχετε να σχολιάσετε, ξεκολουθείτε να έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορθωμένος διάλογος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με το κράτος δικαίου, ε, γιατί ε, από την ε, κυρία Μετσόλα και όλοι οι υπόλοιποι ομιλητέ αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και στο νέο μηχανισμό. Θα ήθελα να εξηγήσω περισσότερο τι προσπαθώ να κάνω, γιατί είπα θα είμαι επικεφαλής του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρουσιάσουμε και την πρώτη έκθεση φέτος. Καταρχήν, δεν θέλουμε να έχουμε μόνο ένα εργαλείο, ένα μόνο μέσο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και με άλλα εργαλεία όπως το άρθρο Όμως θα προσθέσουμε ένα νέο εργαλείο, το μηχανισμό της ετήσιας έκθεσης. Η ετήσια έκθεση θα είναι ίσως η πρώτη ευκαιρία να οργανώσουμε μια διαδικασία η οποία δεν θα εισάγει διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Θα είναι μια έκθεση που θα αφορά και τα 27 κράτη-μέλη και δεν θέλω να επανέλθω στη συζήτηση για συγκεκριμένα το είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια. Και είχαμε και την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να τα συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Τώρα, ποιο, ήταν το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ήταν η πρώτη ερώτηση. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα στείλω μια επιστολή σε όλα τα κράτη-μέλη για να συστήσουν ένα σημείο επαφής ε, σε όλα τα κρατημέλη προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους τη μελλοντική έκθεση. Όχι γιατί θέλουμε να λάβουμε στοιχεία μόνο από τα κράτη-μέλη. Ε, και με τους οργανισμούς ε, όπως η ΦΡΑ ή με την Επιτροπή της Βενετίας και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να έχουμε την ευκαιρία να εκπονήσουμε την εκθεσή μας. Και ήδη έχουμε πολλά εργαλεία στην Κομισιόν, με το σχάρι, ε, το scoreboard, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη. Έτσι, λοιπόν, ε, θα έχουμε τις πρώτες συναντήσεις με τα κράτη-μέλη το Φεβρουάριο και φυσικά θα ενημερώσω το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ίσως για την πρόοδο που θα σημειώσουμε για την εκπόνηση της έκθεσης. Το πλαίσιο. Τι είναι σημαντικό. Πρέπει να αναφέρουμε τα πρότυπα σε μια τέτοια έκθεση. Ποια είναι τα εφαρμοστέα πρότυπα σε διάφορους τομείς και θα το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι έχουμε κάποια πρότυπα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή και από άλλους οργανισμούς και επίση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι σαφέ γιατί θέλω να επιβεβαιώσω ε, για το ότι πρέπει να εφαρμόσει η Κομισιόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θα έχουμε καταρχήν τον ε, προσδιορισμό των προτύπων, κατόπιν θα περιγραφεί η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και κατόπιν ε, θα παρουσιάσουμε τις κινήσεις που έχουν εντοπιστεί στα διάφορα κράτη-μέλη και φυσικά θα έχουμε και τις συστάσεις. Τώρα, ποια είναι τα θέματα που θα εξετάσουμε. Την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο. είναι το πρώτο στοιχείο του κράτους δικαιού. Πρέπει να έχεις ανεξάρτητα δικαστήρια προκειμένου να μπορέσεις ε, να απολαύσεις ως πολίτης τα δικαιώματά σου. Και ε, επίση ένα δεύτερο θέμα είναι η διαφθορά. Άκουσα πολλές ερωτήσεις για τη διαφθορά και τις εγκληματικέ οργανώσεις. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά επ' και όχι μόνο στον μηχανισμό, αλλά και με άλλα εργαλεία δικαστική συνεργασία. Όμω αυτό θα είναι σημαντικό κεφάλαιο του μηχανισμού στην έκθεση. Τρίτο στοιχείο είναι η πολυφωνία των μέσων μαζική ενημέρωση και εκεί θα δούμε αν χρειαστεί να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία και άλλα ζητήματα. Για να κάνουμε τι, για να έχουμε μια πρώτη έκθεση θα έχει ευρύ πεδίο εφαρμογή, αλλά ίσω δεν θα θέλουμε να καλύψουμε όλα τα πιθανά ζητήματα στην πρώτη έκθεση και θα έχουμε και άλλα εργαλεία για να καλύψουμε άλλου είδους στοιχεία. Να αναφέρω ένα, θα έχουμε το χάρη συγκεκριμένη έκθεση για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ίσως θα έχουμε μια έκθεση που θα έρχεται από την Κομισιόν για τη Δημοκρατία. Τελικά λοιπόν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα, όμως θέλουμε να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα και όχι μόνο την εξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά θα περιγράψουμε την κατάσταση σε όλα στα κράτη μέλη και θα αναλύσουμε τους κινδύνους, όπως σας είπα και θα έχουμε και συστάσεις για να κάνουμε τι. Καταρχήν, να ανταλλάξουμε τις βαλτιστικές πρακτικές και να έχουμε και ένα προληπτικό ρόλο. Είναι δυνατόν ε, να βελτιώσουμε τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πείσουμε κάποια μέλη να μετακινηθούν ε, και να θετήσουν καλά πρότυπα σε διαφορούς τομείς. Φυσικά, αν χρειάζεται, θα είναι ένα καλό εργαλείο προκειμένου να εισαχθούν διαδικασίε σε παραβάση, αν είναι η μόνη λύση για την Κομισιόν. Σω θα είναι για ένα καλό μέσο για να κάνουμε άλλε συζητήσει. Ξέρω ότι έχουμε συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και την πιθανή ερωσιμότητα. Σε ποια βάση. Ίσως στη βάση μια τέτοια ε, έκθεση με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία όπου θα αναλυθεί το κράτος δικαίου. ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και σε άλλους τομείς. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές αποδείξεις, αλλά ξέρω ότι κάνετε κάποιες συζητήσει ε, στο θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων σχέση με το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Ίσως η έκθεση αποτελεί ένα ε, καλό σημείο συζήτησης. Ίσως ε, λοιπόν στην έναρξη της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την έκθεση και να έχουμε πραγματική συζήτηση επί της έκθεσης στο πλαίσιο του διαλόγου που θα οργανωθεί κατά τη Γερμανική Προεδρία. Φυσικά, η έκθεση είναι μια έκθεση της ε, Κομισιόν. Ε, θα πάει στο Συμβούλιο, αν το Συμβούλιο θέλει να οργανώσει πολιτική συζήτηση με αξιολόγηση ομοτήμων σε επίπεδο κρατών μελών ε, και Επίσης θα έρθει και στο Κοινοβούλιο και από εσά εξαρτάται να οργανώσετε επίσης μια συζήτηση για την έκθεση αυτή και ίσως και για άλλα στοιχεία είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί είναι ο καλύτερος ε, τρόπος ε, τελικά να έχουμε την ε, ίδια διαδικασία για τα πολιτικά κριτήρια της ενωσής μας, για τις αξίες μας, που έχουμε για την δημοσιονομική κατάσταση και για τη διαδικασία σύγκλησης στις διάφορες οικονομίες των κρατών μελών. Και είμαι βέβαιος ότι Ήρθε ο καιρό να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πολλέ συζητήσει στο παρελθόν, αλλά φέτο θα έχουμε τη δημοσίευση τέτοια έκθεση. Και πάλι, έχουμε όλα τα εργαλεία, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν και τα άλλα εργαλεία, το άρθρο 7, αλλά και τη διαδικασία επί παραβάση και άλλα εργαλεία για να προωθήσουμε την κουλτούρα του κράτους δικαίου στα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό γιατί ίσω ε, το πιο σημαντικό στοιχείο για το κράτο του είναι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία και να έχουμε μια πολιτική συζήτηση για τι ε, αξίε μα ε, και για το άρθρο 2 τη συνθήκη. Κάτι δεύτερο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Συγγελία. Άκουσα πολλά σχόλια. Καταρχήν, ε, στα τέλη του έτους θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Νοέμβριο του 2020 είναι ο στόχος που έχουμε θέσει. Έχουμε την κυρία Κέβεση που είναι επικεφαλής εισαγγελέα. Ε, προσπαθούμε ε, να έχουμε και ένα σώμα. Θα πρέπει να πείσω ένα κράτος μέλος για να έχουμε τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να ληφθεί απόφαση. Και κατόπιν θα αναλύσουμε την δημοσιονομική κατάσταση έχω λάβει τα στοιχεία του προπολογισμού, τα δεδομένα του προπολογισμού του προηγούμενη Κομισιόν και θα έχετε δει στην πρόταση τη προηγούμενη Κομισιόν για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο κάποια στοιχεία για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν καινούργιε συζητήσει για το θέμα αυτό, γιατί ε, υπάρχουν νέε αξιολογήσει για τον αριθμό των ε, που έρχονται ε, ε, από τα κρατη email. Θα τα λύσω αυτά με την κυρία Κέβεση και επίση ε, θα ζητήσω από την κυρία Κέβεση να απευθυνθεί σε εσά, αλλά να πάει και στο Συμβούλιο και να εξηγήσει τι νέε αξιολογήσει για τον προπολογισμό, αν χρειαστεί. Φυσικά θα ζητήσουμε αύξηση του προπολογισμού στι συζητήσει για το πολιτεστικό συνομικό πλαίσιο. Αλλά καταρχήν θέλω να λάβω όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία. Έχω ένα πρώτο έγγραφο, αλλά θα ήθελα ε, διευκρινήσει που να έρθουν από το προσωπικό για την κυρία Κέβεση και κατόπιν ε, θα δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Ε, και πριν είδα και το διευθυντή της Eurojust εδώ στην επιτροπή σας και αν υπάρχουν κάποιες αιτήσει, κάποια αιτήματα από την Eurojust, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη δικαστική συνεργασία, ε, στην Ευρώπη, αν χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερο προπολογισμό για τη Eurojust και αυτή την κατάσταση θα την αναλύσουμε. Γιατί έχω λάβει μία πρόταση από την προηγούμενη Κομισιόν και πάλι για τους οργανισμούς και για τη Eurojust. Ξέρω ότι υπάρχει μείωση του προπολογισμού στη νέα πρόταση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Όμως και πάλι είμαι ανοιχτό να συζητήσω με τη Eurojust και θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη παρουσία στις κατάστασης και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο λιγμών στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αλλά φυσικά έχουμε αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή που προέρχονται από μια απόφαση από το Μάιο του 2019. Επίση, ε, θα είναι δυνατόν να έχουμε ανοιχτή συζήτηση με τη Eurojust για το θέμα αυτό. Τώρα, για το Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων, GDPR. Είπα από την αρχή ότι θέλουμε να έχουμε ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές για να εφαρμόσουν σωστά και ομοιόμορφα τον GDPR σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι δυνατό λοιπόν να δώσουμε υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη, σε ανθρώπινους πόρους για να γίνει αυτό στα κρατημέλια, φυσικά στο τέλος της διαδικασίας είναι επίσης δυνατόν να εισαγάγουμε κάποιες διαδικασίες επί παραβάση. Έχουμε και ε, την ικανότητα να βοηθήσουμε αν είναι δυνατό και αν έχουμε καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και αν όχι, ίσως είναι το καθήκον μας ε, να προσφύγουμε στο δικαστήριο και να ζητήσουμε καλύτερη εφαρμογή όλων των στοιχείων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε καλύτερη εφαρμογή για τους πολίτες γενικά. Είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ καλός ο κανονισμός, όμως δεν είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιείται ο κανονισμός ε, από όλους τους πολίτες με πλουστευμένο τρόπο. Ίσως με την τεχνητή νοημοσύνη να έχουμε νέες δυνατότητες ε, για να βοηθήσουμε τους πολίτες να εφαρμόσουν σωστά τον κανονισμό και θα συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές στο θέμα αυτό. Ξέρω ότι έχουμε πολλές ε, συζητήσεις ε, για τις εξελίξεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφερθήκατε και σε άλλους τομείς, αλλά καταρχήν για το GDPR. Και αναφέρθηκαν οι βουλευτέ στην κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση και ξέρω ότι είναι σύντομος ο χρόνος για τις διαπραγματεύσεις. Ένας χρόνος δεν αρκεί. Όμως, ε, καταρχήν, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρμόδιο να αποφασίσει ε, για το αν θα σταματήσει η διαπραγματεύση στα τέλη του έτους. Ξέρετε, είναι δυνατό ο Πρωθυπουργό να περάσει νομοθεσία για να παρατείνει το χρόνο. Έτσι λοιπόν εργαζόμαστε σκληρά με τους υπόλοιπους επιτρόπους για να πραγματευτούμε και να αναλύσουμε την κατάσταση και φυσικά θα υπερασπίσουμε μια ορθή εφαρμογή του GDPR. Είπα ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα για τον κόσμο και είμαι σίγουρο ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο σε κάποια άλλη μέρα του κόσμου για την εφαρμογή τη προστασία των δεδομένων. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στον Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα αυτό. Επίση να αναφέρω και τη συζήτηση για τις ηλεκτρονικέ αποδείξει. Δεν θέλω τώρα να επηρεάσω το Κοινοβούλιο, γιατί διαμορφώνει τη θέση του, αλλά εργάζομαι για την διαμόρφωση μια θέση. Είπατε, υπάρχει θέση τη Κομισιόν, είναι αλήθεια, αλλά εγώ τώρα περιμένω συγκεκριμένες προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν και κατόπιν να ξεκινήσουμε τριμερή διάλογο. Είναι αλήθεια, θα προσπαθήσω φυσικά να επηρεάσω και να πείσω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις με ισορροπημένο τρόπο. Ξέρω ότι υπάρχουν ανησυχίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το κράτος δικαίου σε κάποια κράτη-μέλη. Όμως, όπως και για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, αν δεν έχεις προϋπολογισμό, δεν χρειάζεσαι ρεσιμότητα. Αν δεν έχεις ε, την ικανότητα να εργαστείς ε, για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία με πρόσβαση σε υποδείξει αυτέ σε άλλε χώρε δεν χρειάζεται εξαίρεση βάσει του κράτου δικαίου. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν πρώτα ο νέο μηχανισμό και είμαι σίγουρο ότι είναι σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να, να εργαστούμε πιο σκληρά για την καταπολέμηση τη διαφθορά, του οργανωμένου εγκλήματο κτλ. Αλλά το οργανωμένο έγκλημα είναι διασυνοριακή δραστηριότητα. Ξέρετε, στην ομιλία φαινόμενων εσόδων, στη διαφθορά, στο οργανωμένο έγκλημα, αν δεν έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία θα είναι δύσκολο στον πραγματικό κόσμο να εργαστούμε αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ισορροπημένη προσέγγιση και θα εργαστούμε σκληρά. Και θέλω να αναφερθώ στι Ηνωμένε γιατί υπήρχε μια ερώτηση για τι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κλείσω τίποτα με τις ΗΠΑ πριν να υπάρχει εσωτερική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε κοινό όραμα καταρχήν στην Ευρώπη για κατόπιν να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε ε, να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά με άλλου εταίρους. Και είναι αλήθεια ότι όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτη μέρη και με τη ΣΥΠΑ ότι ισχύει αυτό. Είναι ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα. Τώρα, για τη θυματοποίηση. Είδα apply the um, Συγγνώμη, τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, πρέπει ε, να θέσουμε κανόνες για όλα τα θύματα και αν χρειαστεί να αλλάξουμε και κάποιους κανονισμούς. Έχουμε την ε, προσοχή των για τα θύματα τρομοκρατικών υποθέσεων και είναι λογικό γιατί είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουμε και πολλά άλλα θύματα και είναι σημαντικό να οργανώσουμε μια διαδικασία και να έχουμε ένα σύνολο δράσεων και λύσεων για όλα τα θύματα, για τα διάφορα είδη εγκλημάτων. Και μίλησα για τη στρατηγική, δεν είναι για το 2024, είναι από το 2020 μέχρι το 2024, καθ' όλη την περίοδο. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι το 2024 να ξεκινήσω, θα είναι πολύ αργά μάλλον. Μιλάμε για στρατηγική από το 2020 μέχρι το 2024 για τα δικαιώματα των θυμάτων και θα εργαστούμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Για το οργανωμένο έγκλημα για τη διαφθορά κτλ. Είπα, θα είναι σημαντικό τμήμα ε, η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, στον μηχανισμό και στο κράτος δικαίου. Όμως ε, θα εργαστούμε και επί νέων εργαλείων για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους εισαγγελείς στις δράσεις που αναλαμβάνουν κατά του οργανωμένου εγκλήματος της διαφθοράς νομιμοποίησης παρανόμων εισόδων. Και θα προσπαθήσουμε να τοικοποιήσουμε τη συνεργασία και το συνδυασμό αν είναι δυνατόν να έχουμε και καλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως ε, και πάλι δεν θέλω να επηρεάσω υπερβολικά την Επιτροπή σας για τα διάφορα εργαλεία. Ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι ίσως τμήμα της ικανότητάς μας ε, να εργαστούμε για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη. Να επαναλάβω. Θα έχουμε στις 19 Φεβρουαρίου τη Λευκή Βίβλο από την Κομισιόν. Περιμένετε λοιπόν την ανακοίνωση της Επιτροπής πριν απαντήσω τις διάφορες ερωτήσεις. Όμως το δικό μου χαρτοφυλάκιο έχω την ευθύνη να προσπαθήσω να οργανώσω μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλήθεια κύριε Πέτερς, δεν γνωρίζω να υπάρχει οριζόντα προσέγγιση. Θα πρέπει να εργαστώ ε, επί της ικανότητας προστασίας των μηλιών δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων για κάθε πιθανή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να εργαστώ επί της ικανότητας να οργανώσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας ε, για την ασφάλεια των προϊόντων. Έχουμε μια γενική οδηγία και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τέτοια ικανότητα, να έχουμε δίκτυο ασφαλείας για όλε τις διαφορετικές δυνατότητες που θα έχουμε με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο ισχύει για την ευθύνη. Θα πρέπει να εργαστούμε επί του θέματος της ευθύνη και πάλι ίσως να έχουμε ένα κοινό κανόνα για πολλές διαφορετικές δυνατότητες που θα ανακύψουν. Δεν είμαι κατά τις ε, δυνατότητες να έχουμε βέβαια και μια κάρσια προσέγγιση. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα σε κάποιες τομείς ή να οργανώσουμε διαφορετικό τρόπο να προχωρήσουμε. Στην ε, υγειονομική περίθαλψη, το χάρη, ξέρουμε ότι έχουμε ιδιαίτερε περιπτώσει και ίσω χρειάζεται να κάνουμε κάτι, ίσω και στι μεταφορέ και σε άλλου τομεί. Όμω ε, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ μια οριζοντή και μια κάθετη προσέγγισης όμως ε, θα έχουμε μια οριζόντια εγγύηση για όλες τις διαφορετικές δραστηριότητες που θα καλύπτονται. Και θα έχουμε μια λευκή βίβλο. Θα οργανώσουμε λοιπόν διαβουλεύσεις. Και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το θέμα αυτό. Προσπάθησα, Πρόεδρε, να απαντήσω στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη συζήτηση για να επανέλθω στο κράτος δικαίου και στο σχετικό μηχανισμό. Να πω ότι είναι σημαντικό εργαλείο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Αλλά σας παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε πρώτα. Επό άλλο ρόλο, έχω συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια για τη δυνατότητα να έχουμε ε, μια προσέγγιση χωρί διακρίσει απέναντι στα διάφορα κράτη-μέλη, ε, όπω έχουμε και στο δημοσιονομικό, αλλά τώρα θα πρέπει να εργαστούμε Είμαι ανοιχτό να ξανάρθω και να εξηγήσω το προπαρασκευαστικό έργο και το πώς θα προχωρήσουμε, όμως και πάλι θα πρέπει να εργαστούμε. Είμαι σίγουρος λοιπόν θα έχουμε μια έκθεση στο δεύτερο εξάμεινο του έτους, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μια τέτοια έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μετά την παρουσίαση από την Κομισιόν στο δεύτερο εξάμεινο. Έτσι λοιπόν, μέχρι τότε έχουμε προπαρασκευαστικό έργο και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και να απαντήσω σε ένα στοιχείο που αφορά ένα κράτος μέλος. Αποφασίσαμε στο Κομισιόν να ξεκινήσουμε διαδικασία επί παρεβάση για το αίτημα να έχουμε προσωρινά μέτρα για τις πειθαρχικές διαδικασίες στην Πολωνία. Ήταν πολύ σημαντικό και τώρα παρακολουθούμε και τις συζητήσεις στην Πολωνία στο Κοινοβούλιο για το νέο νομοσχέδιο. Όμως είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι σχετικά. Θα αναλύσουμε την τελική εκδοχή του νομοσχεδίου και θα δούμε αν χρειάζεται να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Όμως βλέπω ότι έρχεται και ο πρόσωπος της Κροατικής Προεδρίας, δεν θέλω να με λοιπόν, και φυσικά θα επανέλθω και θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις ε, στην Επιτροπή, ίσως και σε κάποιους τρίμερες διαλόγους. Απλώ θέλω να πω ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο για τα ηλεκτρονικά αποδεκτικά στοιχεία τον επόμενο μήνα. Θα είναι πολύ καλή εξέλιξη. Ευχαριστούμε, ε, Επίτροπε Ρέντερς, και εκτιμούμε πάρα πολύ τις προσπάθειές σας. Ε, συνεχίζεται η συζήτηση με την Επιτροπή μας. Όπως είδατε, είναι μεγάλες οι προσδοκίες και βαρύς ο φόρτος εργασίας και τα εκκρεμή ζητήματα Αναφερθήκατε σε κάποια από αυτά. Το Eurojust που ε, συζητήσαμε το πρωί, ε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό αφορά και επηρεάζει και την εσωτερική ανάλυση του πολιτικού γίγνεσθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη σχέση μας με τρίτες ε, πλευρές, όπως π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Μας θυμά η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Κροατίας και Υπουργού Εσωτερικών που θα μας αναφέρει για την Υπουργική Συνάντηση Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ που έλαβε χώρα στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2019. Καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Κροατικής Κυβέρνησης, κύριο Ντάβορ ε, Μποζίνοβιτς, που εκπροσωπεί την Κροατική Προεδρία. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος κυβέρνησης, αντιπρόεδρος δηλαδή, και υπουργός εσωτερικών. Παραμένει και ο κύριος Ρέντερς που θα λάβει και εκείνο το λόγο για να μας μιλήσει εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Ασφάλεια, προστασία δεδομένων, ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, ε, αμοιβαιότητα σε θέματα θεώρησης, ε, ε, κυβερνοασφάλεια κλπ. Έχουμε προγραμματίσει 45 λεπτά για το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη μέχρι τις 12.30. Έχουμε και συντονιστές όμως μετά και στη συνέχεια απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με παρουσίαση ε, του προγράμματος της ε, Κροατικής Προεδρίας και προτείνω να τηρήσουμε το χρόνο διάγραμμά μας. Θα γίνει ε, συζήτηση με τους συντονιστές και τους υπόλοιπους που θα έχουν επιζήσει από αυτή τη ε, μακρά συνεδρίαση. Παρακαλώ να θυμηθείτε ότι έχουμε συνολικά τρία τέταρτα. Θα ακούσουμε τον κύριο Μποζίνοβιτς και μετά πάλι τον κύριο Ρέντερ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Υπουργέ. Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε την Προεδρία να ενημερώσει την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την έκβαση ε, ε, του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών, Υπουργική Συνάντηση Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ε, που έγινε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Θα σας δώσω μια επισκόπηση των θεμάτων που καλύψαμε σε υπουργικό επίπεδο σε αυτή τη συνάντηση. Όπως γνωρίζετε, συμπρό έδρευε η Φιλανδική Προεδρία, Υπουργό Δικαιοσύνη τη Φιλανδία από εμά και ο Επίτροπο Ρέντορ. Θα δώσω λοιπόν ε, στη συνέχεια το λόγο στον Επίτροπο Ρέντερς για να μπορέσει να σας ενημερώσει και εκείνος ε, για τις επαφές που είχε με τους ομολόγους μας. Όπως ήθιστε, σε αυτού του τύπου διαλόγου με τις Ηνωμένε Πολιτείες η υπουργική διάσκεψη του Δεκεμβρίου έγινε σε εγκάρδιο κλίμα όπου και οι δύο πλευρές ήθελαν ε, να τονίσουν την έντονη δέσμευσή τους για τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης, θέματα κοινού ενδιαφέροντος και μεταξύ αυτών η επιχειρησιακή συνεργασία. Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπήθηκε από τον Γουίλιαμ Μπάρ Υπουργό Δικαιοσύνης και το Τσάτ Βόλφ που εκτελεί χρέη Υπουργού Εσωτερική Ασφάλεια. Ε, βλέπετε σε πόσο υψηλό επίπεδο ε, ήταν η εκπροσώπηση και πόσο σημαντικό θεωρούν οι Αμερικανοί αυτό το διάλογο. Συχνά είναι επιχειρησιακό ο χαρακτήρα του συντονισμού μα, άρα ήταν παρόντε και η Europol και η Eurojust, καθώ επίση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και ο συντονιστής ε, καταπολέμησης τρομοκρατίας. Όπως ε, σίγουρα γνωρίζετε, αυτές οι υπουργικές συναντήσεις δεν έχουν στόχο καμιά διαπραγμάτευση, καμιά συμφωνία για νέα μέσα συνεργασίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μάλλον μια εξαιρετική ευκαιρία να ε, ενημερωνόμαστε και να συζητούμε τα διάφορα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ένα από τα βασικά θέματα φυσικά είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπου και οι δύο πλευρές έχουν μακρά πρακτική συνεργασίας με ορατά αποτελέσματα για την ασφάλεια των πολιτών μας. Επίσης συζητήσαμε τη σημασία ανταλλαγής ε, πληροφοριών για θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας Και επίσης οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πρέπει να δίνουν στοιχεία που παίρνουν από τα πεδία των μαχών και από το PNR και να τα δίνουν στους συνεργάτες στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση, επειδή οι διάφορε ομάδε έχουν διεθνή δράση, θα πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο ε, τι ε, διεθνεί διαπλοκέ ε, και διασυνδέσει αυτών των ομάδων. μάθαμε τι μέτρα έχουν λάβει δύο πλευρές πρόσφατα για να αντιμετωπίσουν ε, τις απειλές στον κυβερνοχώρο ε, και άλλες απειλές ε, ατομικές, βιολογικές, πυρηνικές κλπ. Μη συμβατικών όπλων. Καθώς επίσης και τα συστήματα αεροσκαφών μη επανδρομένων, τα drones. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Και ε, με ειδικές πρωτοβουλίες κοινέ. Η κυβερνοασφάλεια επίσης είναι ένας τομέας υψηλού επίπεδου που χρειάζεται την ειδική προσοχή των διοκτικών αρχών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα η εφαρμογή του δικτύου 5G κινητής τηλεφωνίας συζητήθηκε γιατί συμβαίνονται κίνδυνοι ασφαλείας με αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι ε, αφορά την κατακαιρματισμένη αλυσίδα ε, παροχής ε, υπηρεσιών 5G. Επίσης για την κυβερνοασφάλεια και τον κυβερνοχώρο, οι Υπουργοί σημείωσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ για διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και την αναθεώρηση του δεύτερου πρωτοκόλου της Σύμβασης της Βουδαπέστης για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Επίσης συζήτησαν τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, σε ό,τι αφορά την ε, κρυπτογράφηση από πλευρά των εγκληματιών. και πώς θα βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία ε, των θεμελιδών δικαιωμάτων και στην πρόσβαση ε, των αρμοδίων ε, διοκτικών αρχών σε κρυπτογραφημένα στοιχεία. Άλλο τομέα που υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι οι βρυδικέ απειλές και οι διαδικασίες εκστρατείες παραπληροφόρησης. Αυτά απειλούν την ακαιρεότητα των δημοκρατιών μας. Σημείωσε η διάσκεψη ε, την πρόοδο της ε, πρόσφατης σχετική συνεδρία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για συζήτηση και ανταλλαγή βέλτιστων ε, πληροφοριών για να προστατεύονται οι ελεύθερες και δίκαιε εκλογές. Τέλος, συζητήσαμε ένα θέμα που χρονίζει, που είναι η αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις διαβατηρίων. Εμείς ζητήσαμε να προχωρήσουμε 28 κράτη-μέλη και ΗΠΑ προς την ε, ε, ε, άρση θεώρησης, υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων για την Πολωνία έγινε αυτό. Παραμένουν τέσσερα κράτη-μέλη που χρειάζονται βίζα. γίνονται προσπάθειες να μπουν στο πρόγραμμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Ρέιντερς για να προσθέσει και εκείνο κάποιες σκέψεις σχετικά με την διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν να ακούσουμε τους συντονιστές. Παρακαλώ. Ε, κύριος Ρέιντερς, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω την Κροατική Προεδρία για την εισαγωγή ε, σε σχέση με τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν στην Υπουργική Σύνοδο. Ήταν η πρώτη μου Υπουργική Σύνοδος με βάση τα νέα μου καθήκοντα και οι συζητήσεις έδειξαν νομίζω τη σημασία αυτού του διαλόγου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία και βεβαίως ε, κάποια ζητήματα που μας ανησυχούν από κοινού. Ε, στην ατζέντα για τις απειλές για την ασφάλειά μας ε, μιλήσαμε για μια σειρά από ζητήματα, τη συμφωνία για τους επιβάτες, τον ακραίο εξτρεμισμό της λευκής ακροδεξιάς, το θέμα των ξενομαχητών, την πρόσβαση πληροφορίες και την χρήση ε, των πληροφοριών αυτών στις ποινικέ διαδικασίες. Ε, λειτουργεί καλά η συνεργασία, είναι κάτι που επιτρέπει που βοηθάει και, την, ε, κράτη, και τα κράτη-μέλη και, την, ε, Πολιτείε, ό,τι αφορά τους, επιβάτες καλωσορίζουμε την κοινή αξιολόγηση και εκφράζουμε την ελπίδα ότι η τελική έκθεση θα ολοκληρωθεί σύντομα μετά από τις πληροφορίες βέβαια που θα λάβουμε από τους Αμερικανούς Επίσης συζητήσαμε τον αντίκτυπο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία PNR με τον Καναδά καθώς ε, και την προσπάθεια δημιουργίας ε, παγκόσμιων προτύπων PNR στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, ε Αεροπλοείας. Τόσο ό,τι αφορά τώρα την ακροδεξιά είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ανάγκη, μια, μια ανάγκη καλύτερη κατανόηση τη απειλή. Υπάρχει μια πρόταση η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή ε, από τους συνομοθέτες για τις υβριδικές απειλές ε, έγινε αναφορά στην ε, συνεργασία με τους Αμερικανούς για τα χημική, βιολογική, χημικές, βιολογικές, πυρηνικές απειλές, τα εξεκριτικές ύλες, και βεβαίως τη χρήση των drones, των μη επαδρομένων σκαφών ε, και από τις δύο πλευρές. Ε, για την κυβερνοασφάλεια έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δικτύων και των υποδομών δικτύων 5G και των ενδεχόμενων κινδύνων μεταξύ των οποίων αυτών που συνδέονται με την αλυσίδα διανομής και την, ε, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια ε, πολύ αυστηρή θέση δημοσίως ε, έτσι ώστε να απομακρυνθούν κάποιες επιχειρήσεις από την αλυσίδα διανομής στα πλαίσια του 5G. Ε, από την ευρωπαϊκή πλευρά αναφερθήκαμε στην ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου τη συνολική ε, και την προπαρασκευή βεβαίως των μέτρων μετριασμού και των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου Επικοινωνιών της 3ης Δεκεμβρίου του 2019. Το δεύτερο κομμάτι των συζητήσεων είχε να κάνει με τη δικαιοσύνη στην, στον κυβερνοχώρο. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις πρόσφατα για μια συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση για διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ήταν ένα σημείο κλειδί και για τι δύο πλευρέ. Ε, η Υπουργική Σύνοδο καλωσορίζει την θετική εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Βεβαίω μπορεί να υπάρξει σύναψη συμφωνία μόνο όταν υπάρξει συμφωνία για τους ιστορικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτού νομίζω ότι οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να αναζητήσουν διμερώς με τα κράτη-μέλη λύσεις εφόσον οι διαπραγματεύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ε, καθυστερήσουν. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα παίξει ρόλο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των διμερών συμφωνιών με τα κράτη-μέλη. Ζήτησα από την των ε, διαπραγματεύσεων την Αλεξάνδρα Ζέροφ Σρόντερ να σε ενημερώσει ε, πιο λεπτομερώς για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Οι θέσεις αποκλίνουν βέβαια, αλλά ο στόχος είναι να προχωρήσουμε να βρεθεί κοινό έδαφος, ενδεχόμενο κοινό έδαφος επί και όχι να μπλέξουμε σε μια συζήτηση για τη μορφή που θα πάρει η συμφωνία. Ε, εδώ και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για το δεύτερο επιπρόσθετο πρωτόκολλο στο, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα. Η συζήτηση για την κρυπτογράφηση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Οι Αμερικανοί πιέζουν για να ε, εγκρίνουμε μια σειρά από αρχές που, έχουν που θα ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών να επιτρέπουν πρόσβαση στις αρχές επιβολής του νόμου ε, για, την, για να σπάσει ε, η κρυπτογράφηση ε, σε κάποιες έρευνες. Ε, βεβαίως αυτό δημιουργεί και κάποιες προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου. Ταυτόχρονα πρέπει να, γίνει σεβασ... να γίνουν σεβαστές οι απαιτήσει περί προστασίας ιδιωτικής ζωής. Είναι ένα μέτρο τεχνικό για την προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων. Ε, το να αποδυναμώσουμε την κρυπτογράφηση μπορεί να βάλει και κατά αυτή της προστασία, θα επανέλθουμε με του Αμερικανού στη συζήτηση αυτή, σε μελλοντικέ συζητήσει Ό,τι φορά την ανθεκτικότητα τη εκλογική διαδικασία. είχαμε την πρώτη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων στι 26 Νοεμβρίου του 2019, το καλωσόρισε αυτό η Υπουργική, ε, πρέπει να παραμείνει διάλογο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων ε, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, για το θέμα αυτό. Οι Αμερικανοί επικεντρώνονται κυρίω στην κυβερνοασφάλεια και στις κρίσιμες υποδομές, εξετάζουν όλες ε, τις δυνατότητε παρέμβασης εκεί. Έγιναν συζητήσεις ε, ε, σε θετικό κλίμα και για το θέμα των θεωρήσεων, των θεωρήσεων των αξιωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών περισσότερες πληροφορίες ό,τι αφορά τα ποσοστά άρνησης θεώρησης. Αυτό είναι κάτι που θα οδηγήσει θα βοηθήσει τα κρατημέλη να πάρουν, να δράση πιο εστιασμένα Υπάρχει κοινή δήλωση που ζητάει αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά ε, την, τις θεωρήσεις ε, και την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια προσπάθεια από τους Αμερικανούς ε, γύρω από το ζήτημα αυτό τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στα πλαίσια της επόμενης, της επόμενης τριμερούς συνάντησης. Σε ό,τι αφορά ε, την Πολωνία και την συμμετοχή στο Visa Waiver Program, είπαμε ότι χρειάζεται αμοιβαιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, στα πλαίσια της Υπουργικής Συνόδου είχα μια πρώτη επικοδομητική συζήτηση με το Γενικό Εισαγγελέα, ε, εξήγησα τον νέο, τον νέο μου καθήκοντα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Είχαμε και μια πιο σε βάθος συζήτηση ό,τι αφορά την Αμερικανική προσέγγιση, ό,τι αφορά το ζήτημα της κρυπτογράφησης. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρέντερ σε αμοιβαιότητα. Είναι και αυτό μια αρχή, έτσι. Ε, με τις ΗΠΑ θα ήταν καλό σίγουρα αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, σκεφτείτε το χρόνο για να προλάβουμε. Ξεκινούμε με τους συντονιστές. Έχουμε μισή ώρα. Και είναι και η συνεδρία των συντονιστών. Το απόγευμα, ε, επίσης, ε, η προτεραιότητα, η προτεραιότητα της Προεδρίας. Λοιπόν, από το ΕΛΚ, ο κύριος Μέλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. From the joint ministerial meeting. Σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας για την κοινή υπουργική συνάντηση. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για μια σειρά βασικών τομών που αφορούν την αμοιβή ασφάλεια για τους πολίτες. Η προτεραιότητα για μας είναι κανένα κράτος μέλος ε, να μείνει πίσω στις ε, σχέσεις με τις άλλες χώρες. Επομένως, δεν μπορούμε να δεκτούμε την κατάσταση που πέντε κρατημέλη δέχονται διαφορετική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες συμβιότητες για τις θεωρήσεις ε, για βραχυπρόθεσμα προγράμματα άρση χορήγησης θεωρήσεων Πολωνία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την αναμενόμενη πρόοδο στον τομέα αυτό σε ό,τι αφορά τους ξένους μαχητές, ε, οι Ευρωπαίοι υπήκοοι που ε, συλλαμβάνονται και κρατούνται στις ε, τόπους μάχης από τις ΗΠΑ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, έχουν γίνει συζητήσεις, είχετε βρει έναν τρόπο να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό κατόπιν της κοινή συνάντησης που έλεγε χώρα τον περαισμένο Δεκέμβριο με τη ΣΥΠΑ, σημειώθηκε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών που συλλέγονται σε πεδία μάχης για σκοπούς ε, έρευνας και δίωξης. Θα μπορούσατε να μας πείτε στα πλαίσια ποιας δομής ε, θα γίνει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, ποια βήματα στις διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ ΕΕ έχουν λάβει χώρα καθώς το θέμα συζητάται ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οριστικό κείμενο δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέλο. Να περάσουμε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Μέλο. Δεν ε, χαίρομαι που βλέπω ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τις υπαγιά για τις ηλεκτρονικές ε, και είχαν πει ότι τίποτα δεν θα συμφωνηθεί πριν να έχουμε συμφωνία στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, και ένα από του λόγου είναι ο φόβο ότι μπορεί να δημιουργήσουν, να συνάψουν διμερείς συμφωνίε ε, είπα, όπω έκανε ήδη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να είναι κάποιες ε, συμφωνίε καλές, κάποιες μπορεί να είναι καταστροφή, ισχύει αυτό, όμως ε, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και να αποδυναμώσουμε τα δικά μας πρότυπα για την επιβολή του νόμου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Ξέρουμε ότι η κρυπτογράφηση είναι πολύ σημαντική σε πολλούς ε, τομείς. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ήδη υπάρχουν κάποιες ιδέες ε, για το πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη στα κρυπτογραφημένα συστήματα. Θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση μόνο σε κυβερνήσει και στι δημόσιε αρχέ, είπατε. Αλλά όταν υπάρχει πόρτα, μπορεί η πόρτα αυτή να χρησιμοποιηθεί από πολλού. Έτσι λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε άλλους τρόπους ε, για να λαμβάνουμε τις πληροφορίες αντί να ασχοληθούμε με τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις εκλογές και πώς ε, θα διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές αυτό το κυβέρνο χώρο ότι είναι δίκαιες οι εκλογές. Ανησυχώ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες προκαλεί ανησυχία για τον τρόπο που επιτρέπει στους πολίτες ε, να πάνε στις εκλογές ή τους ε, κρατά μακριά, δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό πρέπει να το έχουμε επίσης κατά νου και σε σχέση με το τι γίνεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και πώς ε, προσπαθούν κάποιοι να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ρινιού, κυρία Ίντβαλτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Πιτροπέ, εκ νέου. Καταρχήν, να πω ότι η ανακοίνωση της κυρίας Φόντερ ότι αυτή η Κομισιόν θα είναι μια γεωπολιτική επιτροπή σημαίνει επίσης ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει κάπως ε, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μια πιο εύρωστη στάση απέναντι στους φίλους μας. Ε, ε, γιατί απέναντι, στην απέναντι Ατλαντικού, γιατί έχουμε μια ιστορία ότι συμπεριφερόμαστε ως υποτελείς. Να ξεκινήσω καταρχήν με το απομένο μου θέμα, το PNR. Είναι προφανές ότι η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ δεν πληρεί σε καμία περίπτωση τα πρότυπα που έχουν τεθεί από την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Κομισιόν λοιπόν υποχρεούται νομικά να θέσει τέλος σε μια συμφωνία που αποτελεί κατάφορη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Κατόπιν, θα ήθελα να δω και κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί για 17 χρόνια τώρα περίπου ακούμε ότι η συμφωνία PNR με τη ΣΥΠΑ είναι ζωτική για την ασφάλεια. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει αποδείξει. Το πρόγραμμα άρση ε, της υποχρεώση θεώρηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αρνούνται ξεκάθαρα να γνωρίσουν ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριφέρονται διαφορετικά, μεταχειρίζονται διαφορετικά τους πολίτες μας. Και ξέρω, τώρα ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να συζητάτε με αυτό, όμω οι προκατοχή σα απλά το δέχονταν αυτό. Φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό να είμαστε φίλοι με του Αμερικανού παρά να υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών μα. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Πρέπει να κάνουν προσπάθεια οι χώρε αυτέ. Όλοι είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Δεν είναι οι Αμερικανοί οι οποίοι θα αποφασίσουν ποια είναι τα δικαιώματά του η Κομισιόν έχει νομική υποχρέωση να καταθέσει πρόταση αναστολής της συμφωνίας και προκατοχώς σας είπε στην Επιτροπή αυτή ότι θα το κάνω αυτό γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Ελπίζω αυτή η Επιτροπή να είναι διαφορετική και να Πράξη το καθήκον τη για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει εγώ ε, να ε, πρέπει ουσιαστικά να με πιέζουν ενώ πρέπει να κάνω το νομοθετικό μου έργο. Ποιοι φίλοι θα σου πούν, Α, θα κάνει αυτό που σου είπα. Διαφορετικά θα σε παρακάψουμε ή θα κάνουμε διμερεί συμφωνίε. Θα ήθελα μια γνωμοδότηση νομική υπηρεσία γι' αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι παραβίαση ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να πει στου Αμερικανού, κοιτάξτε, δεν πραγματευτούμε μαζί σα όταν θα έχουμε οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ε, θα συνάψουμε μόνο μία συμφωνία όταν υπάρχει οδηγία. Δεν μιλάμε εδώ για τη σύνοψη συμφωνία, μιλάμε για τι διαπραγματεύσει. Δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε για τα πρότυπα αν δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και τέλο, Πρόεδρε, έχουμε συμφωνήσει να στείλουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι έχει γίνει για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ε, ΕΜΛΑΤ. Ε, όμως, παρόλο που το ζητήσαμε την επιστολή αυτή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν έχει σταλεί ακόμα. Έτσι, λοιπόν, θέλω να ζητήσω από το δικό σας γραφείο να στείλει την επιστολή και να μας απαντήσει η Κομισιόν. Έχει σταλεί η επιστολή, λέει ο Πρόεδρος. Χτες έμαθα ότι δεν είχε σταλεί. Είναι κάτι πολύ πρόσφατο, μάλλον, αν έχει γίνει. Και περνάμε στον κύριο Μπρέιερ τώρα για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε. αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν ισοδύναμη προστασία θεμελιών δικαιωμάτων με αυτή που επιθυμούμε εμεί εδώ. Μαζική παρακολούθηση, αυτή είναι η πολιτική εκεί. Έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο κατά τη που περιλαμβάνει και βασανιστήρια, περιλαμβάνει ε, ατιμωτικές ε, συμπεριφορές, εκτελέσεις, ε, εξοδικαστικές ε, κρατήσεις, ε, συλλήψεις και κρατήσεις. Είναι λοιπόν θέμα ασφάλειας δικής μας να μην συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς όταν διακυβεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θεμελιώσιτες οι διαφορές. Το να, συνεργαζόμαστε δηλαδή με χώρες που δεν προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο εξαιρετικά, κατ' εξαίρεση και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών. Είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά τη συμφωνία PNR, εδώ έχουμε παραβίαση της απόφασης του δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν μας υποσχέθηκε ότι θα επαναπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Καναδά. Μπορεί να μας επιβεβαιώσετε ότι δεσμεύεστε ε, σε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση και να μας πείτε επίσης ε, τι λένε οι Αμερικανοί γι' αυτό και για το θέμα της κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση αποτελεί, είναι συνώνυμο της ασφάλειας. Αυτό είναι αποτελεσματική κρυπτογράφηση. Είτε μπορεί να έχουμε αποτελεσματική κρυπτογράφηση ή είτε μη αποτελεσματική κρυπτογράφηση. Εάν θέλουμε πρόσβαση από τις αρχές υποβολής του νόμου, θα δώσουμε πρόσβαση ε, και στους hackers και σε τρίτες χώρες έτσι είναι. Με τον ίδιο, από τον ίδιο δρόμο θα περάσουν. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή θεμητή πρόσβαση και να ε, αποκλείσουμε τη μη θεμητή πρόσβαση. Αυτό είναι και το νόημα της κρυπτογράφησης. Ε, να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, κανείς ο οποίος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Δεν το επιτρέπεται να έχει πρόσβαση. Οπότε θέλει προσο... προσοχή, διότι αν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα πει ότι δεν είναι κρυπτογραφημένα. Επίσης διαβάζω παντού επιβολή του νόμου, επιβολή του νόμου, αλλά δεν βλέπω πουθενά τον όρο θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, πρέπει εξίσου ε, σε πρώτη, στην πρώτη γραμμή να είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Ε, αναμένουμε τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα και στη Washington. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρέιερ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος από το ID ούτε από το ECR. Πάμε απευθεία στην Γκουε, η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θέλω να πω το εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι είστε θεματοφύλακα των δικών μας συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, υπάρχει μια αμυδρή διαφορά και παρακαλώ να τη σέβεστε, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε μπερδευτεί λίγο. Το λέω έτσι κάπως κοινικά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Έτσι. Τι να κάνουμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. δεν έχουν ειδικό καθεστώς για τους ε, πολίτες τους ε, από ό,τι για άλλους πολίτες, είτε μ' αρέσει είτε όχι, είναι χαμηλότερο το επίπεδο προστασίας από ό,τι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι η προστασία των δεδομένων στην Αμερική έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών. Εκεί το έχουν εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Ε, και είναι συστηματικό και θα πρέπει να το λύσουμε. Και θα, θέλω να μας προειδοποιήσω όλους να προστατεύουμε τις δικές μας συνθήκες και τη δική μας προστασία των δεδομένων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν δεν το κάνουμε και σοβαρά, τότε δεν ξέρω τι μου γίνεται και πού βρισκόμαστε. Το Privacy Shield, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι, καταργήθηκε. Παρά τις κριτικές και την καταβεκραυγή που υπήρχε και στο Κοινοβούλιο. Και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα το ξανακοιτάξει. Είπαν ότι χρειάζονται και βελτιώσεις για αυτό το σύστημα προστασίας της προσωπικής ζωής. Το συζητήσατε αυτό εκεί στον καφέ που ήπιατε. Θα κάνετε κάποιες βελτιώσεις. PNR με τον Καναδά. Λίστες με τα στοιχεία των επιβατών. Αν δούμε ποια είναι η συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τι αναμένεται, είναι πολύ χειρότερη από εκείνη με τον Καναδά. Και έχουν γίνει αλλαγές. Αυτό τι επιπτώσεις θα έχει. Δεν προτίθεστε καθόλου να το συζητήσετε. Πώς θα προχωρήσετε, προθεσμία καμία θα ακούσουμε. Ποιες είναι οι ε, προσδοκίες σας. Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία με τη ΣΥΠΑ, όπως και να είναι, διμερεί, καλά αυτά είναι ανέκδοτα. Δεν μπορώ παρά να σας πω ε, ότι υποστηρίζω αυτά που προτείνουν οι συνάδελφοι. Και πρέπει να σας πω ότι έτσι που μας τα παρουσιάσετε ανησυχώ πάρα πολύ ε, ε, ε τις δικές μας ε, συνθήκες πρέπει να προστατεύεται, όχι τις αμερικανικές. Πραγματικά μου έχουν σηκωθεί τρέχες κεφαλής με αυτά που ακούω. Μάλιστα, πρέπει να υπάρξει χρόνος ε, και για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και για τον επίτροπο να, να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, ένα λεπτό υπόμενο μιλητής, ο κύριος Πρέσλερ. Ναι, θα, ήθελα να μιλήσω αγγλικά, ευχαριστήσω και τον Υπουργό και τον Επίτροπο. Βουλγαρικά, θα, κροατικά θα μιλήσω Ξέρετε ότι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία είναι οι χώρε οι οποίε δεν έχουν ακόμα, δεν χαίρουν τη αμοιβαιότητα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανισότητα, υπάρχει διάκριση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ένωσης. Βεβαίως, ε, μεγάλο μέρος της δουλειά ό,τι αφορά το σύστημα ε, απαλλαγής αποθεώρησης ε, έχει να κάνει με το ίδιο το κράτος μέλος και πρέπει τα κράτη-μέλη να γίνουν και αποτελεσματικά για να απαντήσουν ε, στα, στα αιτήματα των Αμερικανικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως τι κάνει, πώς η, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσουν να τύχουν απαλλαγής από θεώρηση ε, και τι βλέπετε να μπορεί να συμβεί στο μέλλον γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα να ξέρω γιατί ξεκινάτε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά αποκλειτικά στοιχεία που δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία εμείς εδώ, λέει η κυρία Ντάλη. Ε, και κάποιοι λένε ότι δεν το χρειαζόμαστε και καθόλου. Ε, διότι ουσιαστικά η όποια προστασία των δικαιωμάτων θα πληγεί εδώ. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνα, ε, διασυνοριακή πρόσβαση. Ούτε αυτό δεν έχουμε αξιολογήσει. Οι Αμερικανικέ εταιρείε ε, ήδη έχουν μαζική πρόσβαση στα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών μέσω των, των υπάρχοντων ε, μέσων, ε, μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών και βεβαίω οι Αμερικανικέ εταιρείε είναι που το κινούν όλο αυτό το θέμα από την αρχή. Γιατί λοιπόν λέτε ότι πρέπει, είναι απαραίτητο να φτάσετε σε συμφωνία για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν. Είναι ένας τρόπος ε, τελικά να περάσετε από την πίσω πόρτα επιζήμια, ε, επιζήμιους κανόνες πριν καν εγκριθούν από το κοινοβούλιο αυτό. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο προηγούμενο. Ευχαριστώ. Έχουμε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο κύριος Μπασινόβη καταρχήν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις. Γιατί έχουμε ερωτήσεις που δεν μπορούσαμε να τις ομαδοποιήσουμε. Κάποιος ανέφερε τη Συμφωνία Πιενάρια Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Δεν συζητήθηκε η συμφωνία αυτή στη συνάντηση. Επικεντρωθήκαμε στο πώς να βελτιώσουμε την συμφωνία PNR με τις ΗΠΑ που πρόσφατα αυτόματα ανανεώθηκε για μια επταετή περίοδο και οι δύο πλευρές ανέφεραν τη σημασία της ολοκλήρωσης ε, της αξιολόγησης της ε, λειτουργίας της συμφωνίας ε, PNR και η Κομισιόν σίγουρα είναι σε καλύτερη θέση να δώσει συγκεκριμένε πληροφορίες για τις σχετικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις. Μιλώ εκ μέρους της Προεδρίας αν μιλούσα εκ μέρου τη χώρα μου, θα μπορούσα, χώρας μου, μπορούσα παρά να συμφωνήσω. Αλλά πρέπει να παραδεκτώ ότι και ο Επίτροπο και η Προεδρία ήταν σαφής στο να δηλώσουν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό, θα πρέπει να επιτρέψει ε, ως μέτρο αμοιβαιότητας ε, η Αμερική την ε, δυνατότητα να ταξιδεύουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς θεώρηση και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία υποφελείται από την μη υποχρέωση έκδοση θεώρηση, αλλά δεν δίνει την ίδια δυνατότητα και στα 27 κράτη-μέλη. Επίση, καλέσαμε για μια διαφανή διαδικασία σε ό,τι αφορά το ορόσημα για το πρόγραμμα άρση υποχρέωση θεώρηση και περιμένουμε ο τριμερής διάλογος να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προσχώρηση της Πολωνίας ε, στο πρόγραμμα είναι καλό σημάδι αλλά δεν αρκεί. Η Προεδρία μαζί με την Επιτροπή θα συνεχίσουν να θέτουν το θέμα αυτό στις μελλοντικέ συναντήσεις ε, με τους ε, εταίρους των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ε, για πολύ καιρό την ανάγκη για πού αποτελεσματικό εργαλείο που να επιτρέπει την ε, άμεση πρόσβαση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ε, σε παρόχους υπηρεσιών για την χορήγηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό οδήγησε το Συμβούλιο στο να επιτρέψει πέρσι την έναξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και διόρισε την Κομισιόν ως επικεφαλής διαπραγματευτή. Ίσως η Επιτροπή θα ήθελε να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Όμως, ένα είναι βέβαιο. Η τελική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να είναι συμβατή και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές, για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που είναι διαπραγμάτευση και ε, με το Cloud Act, τον είπα, και θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα, για την αμοιβαία νομική συνδρομή και τη Συμφωνία Ομπρέλα για την προστασία των δεδομένων. Αν μου επιτρέπετε, η Υπουργική Διάσκεψη δεν κατέληξε σε συμπεράσματα για το θέμα της κρυπτογράφησης. Αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία συζήτησης ε, για την κρυπτογράφηση και τις συζητήσεις που συνεχίζονται. Είναι δύσκολο το θέμα για όλους μας, όμως ε, χρειάζεται διεθνή συντονισμένη δράση αν πρόκειται να αναπτύξουμε ένα σύστημα που να διασφαλίζει νόμιμη πρόσβαση των διοκτικών αρχών σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Και αναφέρθηκε και το θέμα των ξένων μαχητών. Έχουμε μία συνεχιζόμενη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα αυτό. Συζήτησαν και οι δύο πλευρές το πώς θα ενισχύσουν τη συνεργασία, κυρίως μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και πώς θα βελτιώσουν το ρόλο των ευρωπαϊκών οργανισμών ε, με την ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα στο Ζάγκρεπ, την Πέμπτη, θα είναι παρόν, παρούσα η επιτροπή μα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων. Θα ξαναδούμε όμω τον κύριο Μποζίνοβιτ, ε, μια και θα παρουσιάσει τις, προ... τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά του ζητήματα εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 27 Ιανουαρίου αν δεν κάνω λάθος έτσι δεν είναι ναι στην επόμενη συνεδρίαση η επόμενη συνεδρίαση των ΗΠΑ θα λάβει χώρα στην Κροατία τον Μάιο ε, στο Ντουμπρόβνικ πολύ ωραία ε, το λόγο έχει η Κομισιόν πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη σήμερα το πρωί. Εμείς θα έχουμε συνεδρίαση συντονιστών και μετά το απόγευμα ξανά εδώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Αντιπρόεδρος για τους ξένους μαχητές. Ε, ε, είπαμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η Europol. η οποία έχει και αυτή υποβάλει σχετικό έτοιμο. Καλό είναι, να, έτοιμο. Καλό είναι να έχουμε ένα διάλογο δύο φορέ το χρόνο με του Αμερικανού. Είναι χρήσιμο και το θέμα τη προστασία δεδομένων προσπαθούμε εδώ και καιρό. Και η προηγούμενη Κομισιόν προσπάθησε να πείσει του Αμερικανού εταίρου ότι είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδο γι' αυτό. Και θα είδατε ενδεχομένω την τελευταία πρόταση στην Καλιφόρνια. Ε, ίσως ενδεχομένως ε, ε, και αλλού. Ίσως και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Είχαμε συζητήσει με τους Αμερικανούς ε, για το θέμα αυτό, για το PNR, αλλά δεν θέλουμε να κλείσουμε, να φτάσουμε σε καμιά συμφωνία, να φτάσουμε σε συμφωνία εμεί ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για, το για τις ε, ηλεκτρονικά πολιτικά στοιχεία. Θέλουμε όμω να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος για να υπάρξει μια πρόταση στο ιστορικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να αλλάξω τη θέση και σε ό,τι αφορά το Privacy Shield, συνεργαζόμαστε βεβαίως ε, ε, λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα την εφαρμόσουμε. Για άλλα ζητήματα, η Συμφωνία PNR Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ετοιμάζει μια αξιολόγηση, μια έκθεση αξιολόγηση, η οποία θα εγκριθεί από το κολέγιο μάλλον τον Απρίλιο φέτο. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει όλη την περίοδο εφαρμογή, από το 2012 δηλαδή έω σήμερα. Η κοινή αξιολόγηση ακολουθεί μια προσέγγιση που αναλύει την προσθέμενη αξία τη επιχειρησιακό επίπεδο αυτή τη συμφωνία και αξιολογεί τα αποτελέσματά τη και τον αντίκτυπό τη. Η αποτελεσματικότητα, η αναγκαιότητα και βεβαίω η αναλογικότητα. Επίση, λαμβάνουμε υπόψη την εξέλιξη του νομικού πλαισίου και της νομολογίας και των δύο πλευρών δεν ήταν στόχος της κοινή αξιολόγησης να αντικαταστήσει τη νέα διαδικασία αναθεώρηση και τους στόχους της. Η ομάδα πάντως αξιολόγησε τη δικλής ασφαλείας και, την, ε, και τους στόχους της αξιολόγησης. Ένα μεγάλος αριθμός νομολογιών, της νομολογίας που εξετάστηκαν για να, επιτευχθεί, αυτοί οι στόχοι της αξιολόγησης. Αντιλαμβάνομαι τα διάφορα σχόλια που έγιναν σε ό,τι αφορά την κρυπτογράφηση. Είναι περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό το λόγο και στις διμερείς συζητήσει με το Γενικό Εισαγγελέα προσπάθησα να καταλάβω ποιες είναι οι προθέσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες για το θέμα αυτό. Θέλω να εξηγήσω λίγο την κατάσταση, τουλάχιστον από δική μας πλευράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η αυξανόμενη χρήση της κρυπτογράφησης από τους εγκληματίες δημιουργεί προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου. Δεν πρόκειται να πάρουμε μέτρα τα οποία θα περιορίσουν ή θα αποδυναμώσουν την κρυπτογράφηση. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πέρα από τα εξυπρακτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στα πλαίσια της ενδέκατης έκθεσης πρόοδου για την ασφάλεια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να αναζητήσει περαιτέρω λύσει. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η εισαγωγή συστηματικών backdoors σε συστήματα ή σε συσκευέ είναι, αποτελεί αποδυνάμωση ε, της ασφάλειας. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν συστημικά backdoors. Ε, εξιολογούμε λοιπόν θέσεις που θα επιτρέψουν εστιασμένες, νόμιμες και αναλογικές δράσεις από τις αρχές υποβολής του νόμου για να βοηθηθεί το έργο της δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της ισχυρής και της προκρυπτογράφησης είναι ένας βασικός παράγοντας για την θέσπιση και τη διατήρηση τη ενιαία ψηφική αγορά, τη προστασία τη ιδιωτική ζωή, των βιβλίων δικαιωμάτων και τη προστασία των δεδομένων των πολιτών. Ζητώνται λύσει για μια πραγματική ανησυχία όμω. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τι αρχέ επιβολή του νόμου να έχουν πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα στην καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι είναι ευαίσθητο και λεπτό το ζήτημα αυτό και παραμένει ανοιχτή για την αναζήτηση λύσεων που να είναι αναλογικές, να ε, δικαιολογούνται και να μην αντιβαίνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ισχυρό μηχανισμό διακυβέρνησης που ε, να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Και για το Visa Waiver γνωρίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Το, το είπα και εισαγωγικά. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τον Καναδά και με άλλους δείχνουν ότι απτή πρόοδο προς μια πλήρη αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την απαλλαγή αποθεώρηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεχούς δέσμευσης και ε, διπλωματικών επαφών. Αυτή η προσέγγιση φέρνει αποτελέσματα και με τους Αμερικανούς. Το Νοέμβριο ε, του 2019 η Πολωνία πλέον ε, συμμετέχει στο πρόγραμμα απαλλαγής αποθεώρησης με τους Αμερικανούς. Ε, αυτή η πραγματιστική προσέγγιση, η συνέχιση της δέσμευσης σε δημοτικό επίπεδο είναι ο σωστός δρόμος και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να συζητούμε το ζήτημα αυτό. Ε, όλοι κάνουμε προσπάθειες, ενισχύουμε τις προσπάθειες για να βοηθήσουμε τα τέσσερα κράτη-μέλη που απομένουν για να μπορέσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί δεσμεύονται να δώσουν στα τέσσερα κράτη-μέλη αυτά πρακτικές οδηγίες έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Οι Αμερικανοί δεσμεύονται ε, να δεχθούν τα τέσσερα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα όταν θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις ε, της ε, Αναστολή όλων των εξωτερικών σχέσεων. Δεν θα διστάσουμε να υπάρξει πράξη κατεξοδότηση εφόσον αυτό οδηγήσει σε πρόοδο. όμω το να το κάνουμε αυτό μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, και να επιδεινώσει τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειε μα θα φέρουν αποτέλεσμα και ένα προ ένα τα τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται εκτό ε, θα συμμετάσχουν τελικά στο πρόγραμμα αυτό απαλλαγή θεωρήσεων. Όπω έδειξε και η πρόοδο που σημαίνει με την Πολωνία. Σας ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μπουζίνοβιτ, για τον κύριο Μποζίνοβιτς για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Υπουργική και τον Επίτροπο Ρέιντερ, βέβαια που είναι πάντα στη διάθεσή μα ε, για να μα δώσει εξηγήσει ε, στο μέτρο των δυνατοτήτων του βέβαια και των αντοχών του βέβαια ε, έως το τελευταίο λεπτό της πρωινής συνόδου